liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, versammelte Öffentlichkeit. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, άρχεται η σημερινή συνεδρίαση. Όπως ξέρετε, άλλαξε λίγο η μερίσια διάταξη. Ξεκινάμε με το θέμα επίθεση πληροφοριακά συστήματα και η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου. Είναι ο κύριος Χέλε, λοιπόν, ο οποίος θα λάβει αποκλειστικά τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε πως ε, η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων έχει ορίσει το κυβερνοέγκλημα ως τη μεγαλύτερη ε, εγκληματική δραστηριότητα που απειλεί τις επιχειρήσεις. Η είπα πριν από τέσσερις εβδομάδες ε, ε, δημοσίευσαν ένα νούμερο στο οποίο περιέχονται νούμερα που δεν, ένα έγγραφο στο οποίο περιέχονται νούμερα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για την Ευρώπη και υπολογίζουν πως ε, έχει κοστίσει γύρω στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια ε, πέρυσι η ηλεκτρονική εγκληματικότητα στην χώρα αυτή οπότε μιλάμε για κάτι το οποίο έχει πλέον διαστάσεις ε, και σημασία στην μακροοικονομία και βεβαίως το θέμα αυτό το παρακολουθεί κυρίως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εν βάση περιπτώσει, ήδη από το πρόγραμμα της Χάγης, της Στοκχόλμης το 2009 και 2010 στην ψηφιακή ατζέντα είδαμε το θέμα της ε, ψηφιακής εγκληματικότητας, κυβερνοεγκληματικότητας και Ξέρετε πως κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, νομικά μέσα, διαφορετικά βεβαίως, αλλά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν ε, τιμωρούν καν το κυβέρνο έγκλημα και δεν υπάρχουν νομικά μέσα για την δίωξη του κυβερνού εγκλήματος. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά νομικά κενά και παραθυράκια που οδηγούν στο ότι γίνονται σε αυτές ε, τις χώρες ε, επιθέσεις και οι διαφορετικοί ορισμοί π.χ. των προσωπικών δεδομένων και του τι είναι κυβερνοέγκλημα δημιουργούν προβλήματα ε, τα οποία οδηγούν στο ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη αλλά και επιχειρήσεις απειλούνται από αυτές τις επιθέσεις. Βεβαίως δεν υπάρχουν σύνορα στο διαδίκτυο, οπότε τίθενται πλέον ζητήματα δικαιοδοσίας και βεβαίως τίθεται το ζήτημα γιατί η Κομισιόν ε, με την συμπλήρωση του κανονισμού του Συμβουλίου του 2005 ε, προσπαθεί να συμπληρώσει την ε, κατάσταση αυτή. Κοιτάξτε, θεωρούμε πως δεν ε, αποτελεί επίμαχο θέμα το ότι θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία των ε, αρχών και των αστυνομικών και να πλησιάσουν κάπως ε, οι ποινές, όπως επίσης και οι αξιόπινες εκείνες πράξεις, όπως παραδείγματος χάρη επέμβαση σε δεδομένα και υπολογιστικά συστήματα, το ποιος είναι υπεύθυνο σε περίπτωση νομικών προσώπων, και η ανταλλαγή πληροφοριών. Βεβαίως τα λέω αυτά γιατί όπως είπα δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα όλα τα κράτη-μέλη και ήταν αναγκαίο να καλύψουμε το θέμα αυτό με την οδηγία. Τώρα, η έκθεση αυτή βεβαίως ε, είχε ως αποτέλεσμα ήδη από την απόφαση πλαίσιο να κινητοποιηθούν αρκετά αλλά όπως σας είπα υπάρχουν ακόμα αρκετά νομικά κενά. Οπότε ήρθα σε επαφή με τον κύριο Χολμαέρ ε, που είναι... με, την κυρία Χολμαέρ, με που είναι αρμόδια από την Επιτροπή Λίμπε για αυτό το θέμα, αλλά διαπιστώσαμε πως η κατάσταση είναι τόσο προβληματική γιατί υπάρχει διακομματική ε, συνεννόηση και η Προεδρία του Συμβουλίου αναμένει να ολοκληρώσει εντός του τρέχοντος εξαμήνου, αλλά υπάρχει η άποψη πως πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια ακρόαση για να ακούσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οπότε είναι ακόμα ασαφές ε, το τι είναι το χρονοδιάγραμμα εντός της Επιτροπής Ελευθεριών. Οπότε αναμένουμε κινήσεις από αυτή την επιτροπή, οπότε δεν μπορώ να σας πω τίποτα για το χρονοδιάγραμμα. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά από την άποψη, από τη σκοπιά της δικής μας επιτροπής. Ε, βεβαίως έχουμε ένα νομικό κείμενο, άρα κλασική υπόθεση και δουλειά της Επιτροπής ΛΥΜΕ αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ε, τις απόψεις ε, του τομέα της οικονομίας γιατί είναι πραγματικά κατεπήγον να λάβουν υπόψη τα, να λάβουν μέτρα τα κράτη-μέλη βλέπουμε τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα κενά τα νομικά βλέπετε τις ε, κυβερνοεπιθέσεις στο ETS το σύστημα εμπορίας εκπομπών που οδήγησε πλήρη κατάρρευση του συστήματος και κλείσιμο του συστήματος και μιλάμε ότι ήταν για μια βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής μας και έδειξε άρα πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα το ότι εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, το ότι υπήρχαν διαφορετικά συστήματα και προσβάσεις ασφαλείας σε κάθε χώρα οι λεγόμενες ε, πίσω πόρτες όπου με σχετικά απλό τρόπο μπόρεσαν να παραλύσουν το σύστημα αυτό για 14 ε, ημέρες. Όχι μόνο να το παραλύσουν, αλλά ήταν μια επιτυχής προσπάθεια να κλέψουν άδειες εκατομμυρίων. Δεν πρόκειται απλά για κατάρρευση του συστήματος, αλλά για μια επιτυχή προσπάθεια ε, να κλέψουν άδειες 30 εκατομμυρίων. Σε σύγκριση π.χ. με μια απλή ληστεία τράπεζα έχουμε τελείως νέες διαστάσεις. Οπότε θεωρώ πως ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις οικονομικές ζημίες ε, της ε, κυβερνοεγκληματικότητας, ειδικά ε, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, διαθέτουν κονδύλια και μπορούν να προστατευτούν και ακριβώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζονται και υφίστανται όλο και μεγαλύτερες ζημιές γιατί δεν έχουν και τους πόρους και την πείρα να προστατευτούν επαρκώς. Είναι λοιπόν σημαντικό να παραπέμψουμε στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Όπως σας είπα υπάρχει ήδη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και η ψηφιακή ατσέντα που παρουσίασε πριν από δύο μέρες κυρία Κρούς. Ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι οι πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη ουσία να ενισχυθεί η εντολή της ΕΝΗΣΑ στο πλαίσιο αυτό κάτι το οποίο συμφωνεί και με την τοποθέτηση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ γενικώ για, για την κυβερνοεγκληματικότητα και ξέρετε όπως είπα σε σύγκριση με τις ΙΠΑ δεν έχουμε ένα ενιαίο μέσο και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες στην οικονομία Εμείς δεν έχουμε ευρωπαϊκή εικόνα για το τι σημαίνει αυτό ως ε, οικονομική ζημιά. Οπότε το θέμα είναι πού θα είναι αυτές οι αρμοδιότητες ε, στο μέλλον. Και παρά το ότι δεν θέλουν, ευρωπαϊκά, δεν θέλουν κάποια κράτη-μέλη να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και να πάει παραδείγματο χάρη στην ε, Europol, θα πρέπει να έχουμε κάποιον φορέα ο οποίος θα παρακολουθεί αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια τεχνικά τώρα θέματα τα οποία συζητιούνται ήδη στον ε, κόσμο της οικονομίας Κοίταξε, η πρώτη, άμυνα, η πρώτη γραμμή άμυνας όπως λένε οι Αμερικανοί δεν είναι οι αρχές, η αστυνομία αλλά οι τηλεπικοινωνιακές ε, επιχειρήσεις. Και άρα και στην Ευρώπη ούτε τα κράτη-μέλη είναι αυτά γιατί δεν έχουν ούτως ή άλλως και τα μέσα να το κάνουν. Και πρέπει να αναλύσουμε το εάν ε, οι απειλές ε, που αναγνωρίζονται εδώ πέρα είναι όντως οι απειλές που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Π.χ. δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα botnets που είχαν κάποια μεγάλη σημασία στο παρελθόν για το κυβερνοέγκλημα αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί ειδικά από τον κλάδο που θεωρούν πως τα botnets δεν είναι τόσο πλέον επικίνδυνα αλλά αυτό το οποίο λέμε στοχευμένες επιθέσεις targeted attacks σε συγκεκριμένες ε, υποδομές. Πρέπει λοιπόν να ερευνήσουμε το θέμα και στο πλαίσιο του προγράμματος ε, πλαίσιο για την έρευνα. Όπως σας είπα μας λείπουν τα στατιστικά στοιχεία και θα πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει μια συνέργεια των διαφόρων μέσων που χρησιμοποιούμε σε διαφορά προγράμματα γιατί όπως είπα ασχολούμαστε κυρίως στο πέρασε την εκθέση με την νομική πτυχή οπότε σας ευχαριστώ για την υπομονή σας οπωσδήποτε το θέμα θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια σημαντικό είναι να καταλάβουμε και οι ίδιοι πως δεν έχει νόημα να ακολουθούμε την ε, κοινοβουλευτική τακτική των μικρών ε, φέουδων ε, και ο καθένας στην Επιτροπή του να κάνει διαφορετικές εκθέσεις για το ίδιο θέμα, αλλά και εμείς να συνεργαστούμε με τις άλλες επιτροπές, με την κυρία Χολμάιερ, με την οποία συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά και είναι πραγματικά πάρα πολύ ανοιχτή και δεκτική στην άποψή μας, γιατί θεωρεί πως δεν είναι θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουν μόνο οι κυβερνήσεις ε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εδώ πέρα η συνεισφορά του κλάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτος ο σκιοδησηγητής ο κύριος Έντσου. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο σκιώδης εισηγητής για αυτή την έκθεση από την ομάδα των σοσιαλιστών. Ταυτόχρονα τυχαίνει να είμαι ε, σκιώδης εισηγητής και για τη βασική έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Λοιπόν, κυβερνοεπιθέσεις, ε, κυβερνοτρομοκρατία επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικής ε, κατά ε, κυβερνητικών θεσμών ή θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η τάση που παρατηρείται. Ως συνομοθέτες ε, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της ευρωπαικης ενωσης αυτη ειναι η ταση που παρατηρειται Όσοι αιτίας του φαινομένου. Στην αλήθεια Ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και εγώ θα ήθελα να δείξουμε ιδιαίτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων κυβερνοεγκληματικότητας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις εσκεμμένες και τις μη εσκεμμένες επιθέσεις γιατί είναι σημαντικότατε οι κυρώσεις που θα προβλέπονται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του ποινικού δικαίου, ενισχυμένη εναρμόνιση θα έλεγα, γιατί είναι διασυνοριακό το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το αναδυόμενο φαινόμενο από μόνα τους και ε, θα απέθυνα την εξή έκκληση. Οι ειδικευμένοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπω η Europol και η Eurojust θα πρέπει να επιληθούν ε, του ζητήματο. Επίση θα πρέπει ε, να προβλεφθούν κυρώσει για την παράνομη υποκλοπή συστημάτων πληροφορικής και άλλες, άλλου είδους επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Προ το παρόν ε, αυτό που υπάρχει είναι συντονισμός ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών. Θα πρέπει να ε, κυκλοφορούν καλύτερα οι πληροφορίες ε, για τις διάφορες επιθέσεις που σημειώνονται. Ε, άρα θα χρειαστεί σημείο επαφής σε κάθε κράτος μελός ούτως ώστε να καταγράφονται αμελητή και με αποτελεσματικό τρόπο όλες οι επιθέσεις. Τώρα, η οδηγία για τις επιθέσεις κατά των πληροφορικών συστημάτων θα δώσει ένα χειρό μήνυμα για τους κυβερνοεγκληματίες και τους hackers. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Προστασία των Υποδομών και των Δικτύων βασίζεται σε πέντε διαφορετικούς πυλώνες. Πρόληψη, αναγνώριση των φαινομένων, ε, ε, ε, άμβλυνση των φαινομένων και ούτω καθεξής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής ανέφερε ότι μόνο 12 κράτη-μέλη έχουν οργανώσει ασκήσεις μεγάλης κλίμακος για θέματα ασφαλείας ε, για την ε, διόρθωση και επανόρθωση των ζημιών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, το ταχύτερο δυνατό να μεταφέρουν στην νομοθεσία τους τα σχετικά μέτρα ε, και να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές δικαστικές αρχές ε, για την παράνομη παρέμβαση και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής. Από βιομηχανικής πλευράς οι κυρώσεις ε, για, κατά των εγκληματιών ε, για τις παράνομες ε, παραμβολές θα μας οδηγήσει σε προστασία των βιομηχανιών, των μεγάλων εταιριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βασίζονται στο πληροφορικό του σύστημα για να είναι βιώσιμες οι εμπορικές τους δραστηριότητες. Επίση, παραπέμπω στη Σύμβαση του 2001. Θα πρέπει να ε, ξαναρχίσουμε το διάλογο και τις διαπραγματεύσει. Θα είναι μακρές. Η Σύμβαση ήδη ορίζει την ε, απαράνομη πρόσβαση, την υποκλοπή, την ε, παρεμβολή, τι απάτες και τις κυρώσει. Προσβλέπω στην συνεργασία με τον κύριο Έλλερ για την έκθεση αυτή καθώς και στη συνεργασία με τους άλλους και όλους εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσουκαλάς. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που οι συνάδελφοι ανέφεραν ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Νομίζω όμως ότι αυτό που επεσήμανε ο κύριος Έλερ ε, είναι το σημαντικότερο. Είναι όλα σημαντικά ως προς τις ρυθμίσεις το ζήτημα όμως είναι βαθιά τεχνικό. Θα πρέπει να ε, σας πω λίγο από την εμπειρία από τότε που ασκούσα το επάγγελμα του καθηγητή διδάσκαμε στα ακροατήρια ότι σύμφωνα με τον ορισμό η πληροφορία έχει τις εξής ιδιότητες. Έχει την ιδιότητα να αποθηκεύεται, να διαδίδεται, να ανακτάται και να αναπαράγεται να επιδέχεται μετατροπή και φαλκίδευση και να πολλαπλασιάζεται. Εάν αυτό το συνδυάσετε με την σύγκληση των τεχνολογιών πληροφορικής σε σχέση με την δικτυακή τους επικοινωνία και κάνοντας χρήση και του κανόνα της λογικής που λέει οτιδήποτε περνάει από ένα μυαλό για να υπάρχει θα υπάρξει, θα περάσει και από ένα δεύτερο ο αγώνας εναντίον της κυβερνοτρομοκρατίας ή των κυβερνοεπιθέσεων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιληθεί, όπως είπε ο κύριος Έλερ, με έρευνα επί του αντικειμένου. Είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα που έχει μεγάλη σημασία. Θα σας θυμίσω από το 1985 ο Άλβιν Τέφλερ στο βιβλίο του «Το τρίτο κύμα» υποστηρίζει ότι η μελλοντική τρομοκρατία θα είναι η δικτυακή τρομοκρατία για κάθε δίκτυο κάθε μορφής. Φτάσαμε τώρα να επαληθεύεται αυτό και το ζήτημα αν είναι σοβαρό για την άσκηση της εξουσίας των κρατών εξίσου σοβαρό όπως είπε ο κύριος Έλερ και για την οικονομία, τη βιομηχανία και την ε, επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό θα έπρεπε, ακούω με ευχαρίστηση ότι τα κείμενα αυτά ε, παίρνουν όλες τις πρόνοιες. Ε, δέχομαι ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τον Ενίζα και θα έπρεπε να τον ενισχύσουμε με τεχνικά μέσα καθώς και την έρευνά μας για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σέλερ ξανά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Βλέπω οι βασικιώδεις και οι συνάδελφοι γνωρίζουν το θέμα και αυτό είναι αναγκαίο γιατί είχαμε πολλές αλλά κατακαιρματισμένες προσεγγίσεις στο παρελθόν. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που μας αφορά και τους ίδιους. Ε, ξέρετε πως ε, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προστατευόμαστε για το ότι δεν έχουμε παντού wireless LAN. Οπότε δεν είμαστε γι' αυτό το λόγο τόσο ευάλωτοι επιθέσεις. Αλλά δεν είναι λύση αυτή, αν και είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό το οποίο μου φαίνεται ενδιαφέρον εδώ πέρα, όσον αφορά την αναρμόνιση του δικαίου, είναι και αυτή βεβαίω μια επιτυχία, αλλά πρέπει να δούμε γενικότερα την προσέγγιση μας. Πάρα πολλές από τις ε, πράξεις οποίες θέλουμε να κάνουμε αξιόπινες δεν έχουν καν ε, οριστεί. Κάθε μέρα λαμβάνουμε νέες πληροφορίες για τρόπους ε, δράσης οι οποίες βεβαίως προκαλούν βλάβη σε άτομα, Ευρωπαίους πολίτες, επιχειρήσεις αλλά δεν καλύπτονται από τις νομικές έννοιες και εάν για να αντιληφθείτε τη διάσταση, αν ρωτήσετε σήμερα τον κύριο Μπαρόσο, την κυρία Κρούς την κυρία Μάλμστρομ, αν τους ρωτήσουμε, είναι η σημερινή ημέρα επικίνδυνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική ασφάλεια ή όχι. σε αντίθεση με κάποια κράτη-μέλη ή της ΕΠΑ δεν θα έχετε απάντηση για το αν έχουμε κάποια ένταση αυτής της δραστηριότητας ή όχι. Δεν έχουμε δηλαδή μια εικόνα. Και θεωρώ άρα πως είναι σημαντικό όταν μιλάμε για εναρμόνιση του δικαίου να είναι σαφές πως ε, πολλά από τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αξιόπινες πράξεις είναι τόσο καινούρια ώστε και στα κάτω εκείνα τα οποία υπάρχει νομικό πλαίσιο καλύπτονται μόνο εν μέρη και αυτό σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να δούμε ευρύτερα το ζήτημα χρειαζόμαστε επιγόντως ισχυρότερη ενίσα, επιγόντως Ε, όχι μόνο να μιλάμε για προδιαγραφές, χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, ισχυρότερη ενίσα, χρειαζόμαστε ευρύτερη προσέγγιση. Π.χ. στη ΣΥΠΑ βλέπετε πως ε, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας έχει χιλίους ειδικού, για την ε, κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή μόνο οι δυνατότητες από πλευράς ε, προσωπικού αν τις συγκρίνεται, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε 200 τα άτομα. Και βεβαίως η οικονομική διάσταση δεν είναι μόνο η πλευρά της εγκληματικότητας. Έχουμε ουσιαστικό κίνδυνο. Μιλάμε για την βάση των υποδομών ε, της ε, βιομηχανίας. Ε, το θέμα δε, του συστήματος εκπομπών μας έδειξε πόσο επηρεάζονται και κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές που δεν τις είχαμε καν συνδέσει με το θέμα αυτό και το επαναλαμβάνω γιατί ίσως δεν είναι γνωστό. Ίσως τόσο. Η πλατφόρμα αυτή ε, κατέρευσε, αλλά η προσπάθεια επέτυχε. 30 εκατομμύρια σε άδειες ε, κλάψαν. Πάει, τελείωσε αυτό. Και θα ήθελα να, να σας παρακαλέσω να μην δούμε μόνο το θέμα ως μια έκθεση, αλλά να ζητήσουμε από εδώ και μπρος μονίμως η Κομισιόν να ασχολείται με το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας. Και οι περιορισμοί λόγω εγωισμών των κρατών μελών πρέπει να σταματήσουν, γιατί δεν υπάρχει πλέον προστασία ενός μόνο κράτους μέλους. γιατί πλέον ε, είμαστε τόσο ισχυροί όσο ο, ασθενό, ο ασθενέστερος κρίκος στην ε, Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το προωθήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση. 11 ε, Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για τροπολογίες. Αυτό σχετίζεται βέβαια με την ΛΥΜΠΕ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ανάλυση των ε, επιλογών για μείωση κατά 20% και ο κίνδυνος ε, διαρροής άνθρακα. Λοιπόν, η κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν Σίσελη έχει πρώτο λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, έλαβα 188 τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι συναντήθηκα τακτικά με τους ε, σκεώδεις εισηγητές και θα βρούμε καμιά εικοσαριά συμβιβαστικές τροπολογίες. Όπως ε, θα διαπιστώσατε, και εγώ κατέθεσα τροπολογίες. τροπολογίες οι οποίες θέλουν να καταστήσουν πιο απλό και πιο διαφανές το έγγραφο. Μετά έχουμε αυτή, έχουμε την roadmap ε, του 2050 ε, και την ενεργειακή ασφάλεια και επίσης τις τροπολογίες τις οποίες θα προσπαθήσω να σχολιάσω και να τις κατατάξω σε διάφορες ομάδες. Έχουμε προπολογίες οι οποίες κρίνουν τη θετική ή την αρνητική εξέλιξη προς μια κοινωνία και επιπτώσεις προς μια κοινωνία με λιγότερες εκπομπές. Εγώ αυτές δεν τις υποστηρίζω, διότι εγώ θέλω ναι να έχουμε τις αρνητικές ή τις θετικές πτυχές, οικονομική κρίση για παράδειγμα. η οποία ναι μεν μειώνει τις επιπτώσεις των εκπομπών αλλά ταυτόχρονα ε, δημιουργεί και μείωση των επενδύσεων. Μετά έχουμε τις τροπολογίε που αφορούν στο ETS. το οποίο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει κανονικά και αυτό λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη Νέα Ζηλανδία όμως και στην Καλιφόρνια Φαίνεται αυτό το μέτρο να είναι σωστό. Δεν υποστηρίζω εγώ λοιπόν τις τροπολογίες που θέλουν να καταργήσουμε το σύστημα ETS. Ε Δεν θέλω επίσης να υποστηρίξω τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες θέλουν μια ριζική μετατροπή του ETS ε διότι θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πρώτα 100%. Μετά έχουμε και τους στόχους που θα μπορούσαν σίγουρα να είναι πιο φιλόδοξοι άμα είχαμε αντίστοιχες φιλοδοξίες και σχεδιασμούς προς τα έξω και από τις άλλες χώρες. Θεωρώ κατά συνέπεια ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι θετική. Οι αιτιές δεν θα πρέπει να θυχθούν, να... θα πρέπει να προσεγγίσουμε το 20% ενεργειακής αποτελεσματικότητας που σημαίνει 25% μείωση των εκπομπών για το 2020. Ορισμένες τροπολογίες αναφέρονται και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να, σταθούμε, να παραμείνουμε στη θέση της έκθεσης Μπένσεν. Υποστηρίζω τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες μιλάνε για καταβολή μεγαλύτερων προσπαθειών στον τομέα των μεταφορών και των οικοδομών που είναι εκτός του ETS. Ε οι τροπολογίες όμως για την έρευνα είναι άστοχες. Υπάρχουν μετά και άλλες τροπολογίες, είναι οι τροπολογίες εκείνες όπου οι συνάδελφοι παίρνουν θέση γύρω από τις διάφορες τεχνολογίες. Στην πολιτική όμως εμείς πρέπει να θέτουμε πολιτικά κριτήρια αυτό πρέπει να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά οι εμπειρογνώμονες θα είναι αυτοί που θα μας πούνε αυτή η τεχνολογία είναι καλύτερη ή άλλη όχι. Στις μεταφορές το να δεχτούμε την τροπολογία που λέει ότι θα πρέπει να, να στοχεύουμε μόνο στην κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν νομίζω ότι είναι εύστοχο. Μετά έχουμε τροπολογίες σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Αυτό το έγγραφο δεν είναι ένα έγγραφο υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, οπότε δεν στέκει. Μετά έχουμε και άλλες τροπολογίες που καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 36 τροπολογίες τις οποίες υποστηρίζω που καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τα τρέχοντα προγράμματα. Υπάρχουν μετά και οι τροπολογίες που προτείνουν άλλου είδους λύσεις για τη μείωση των εκπομπών και τις οποίες υποστηρίζουν Είναι θετικές προτάσεις. Η Κομισιόν, ας πούμε, θα έπρεπε να θέσει προδιαγραφές για τις μεταφορές, δίκτυα. Αυτά είναι θετικά πράγματα. Μετά υπάρχουν και προτάσεις σχετικά για το ρόλο των TIC για, την, για τις εκπομπές, έχουμε το πρόγραμμα CHIP για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, έχουμε την τροπολογία 122 ας πούμε που είναι πολύ σωστή. Και αυτές τις ε, τροπολογίες τις υποστηρίζω. Μετά μου αρέσουν και οι τροπολογίες εκείνες οι οποίες αναφέρονται στις ΜΜΕ για την υλοποίηση των ε, νέων τεχνολογιών. Η κυρία Χέρτζοκ κατέθεσε σχετικές τροπολογίες και τις υποστηρίζει. Μετά έχουμε τη συνάδελφο Καρβάλιο η οποία λέει για μια τομεακή προσέγγιση. Εγώ συμφωνώ. Σε ορισμένες τροπολογίες υποστηρίζεται ότι μέχρι τώρα τα διάφορα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν έχουν ληφθεί υπόψη και ότι θα πρέπει να τα ξαναδούμε Υπόθηκε ότι στο κείμενο δεν είμαι παρκώς ακριβής. Η τροπολογία 93 που αφορά στην υποδομ... στις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές <coughs> και οι τροπολογίες εκείνες που υποδεικνύουν ότι το αίτημά μου για την ευελιξία των ETS δεν είναι ευστοχή, είναι οι 99, οι 100 και 101 τροπολογίες. Μετά είπαμε έχουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες για αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας Μετά έχουμε και εκείνες ε, τις τροπολογίες που υπογραμμίζουν τη σημασία του CCS και θα ακούσω τώρα τους συναδέλφους. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές για την εξαιρετική τους συνεργασία όπως επίσης και τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με υποστήριξαν ε, και για την έκθεση και για τις ε, τροπολογίες. Αρχίζει η συζήτηση. Ευχαριστώ. σας πω πριν δώσω το λόγο συναδέλφους πως έχουμε φοιτητές ε, από το Ινστιτούτο Μποτσόνη στην Ρέτζιο Καλάμπρια. Ε, σας καλωσορίζω, θα δείτε και πώς συζητάμε εδώ μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Γκρότε. Ναι, χαιρόμαστε για το ότι έχουμε και επισκέψεις και νέους, και νέους ανθρώπους, να δούμε για κανένα νέο. Και ε, συμμετέχει λοιπόν και το κοινό και ελπίζω να αποκομίσουν κάποια πράγματα από αυτό το θέμα. Πρόκειται εδώ πέρα λοιπόν για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Μια έκθεση πρωτοβουλίας Ε, συντάσσεται όταν το δέχεται μια μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το οποίο είδαμε την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να το δούμε αυτό γιατί είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προεργασία εδώ πέρα και η συνάδελφος, η συγγήτρια έκανε πάρα πολύ δουλειά, υπέβαλε αξιόλογες συμβαστικές ε, πρωτοβουλίες που, με συγχωρείτε, τροπολογίες μπορούν να αποτελέσουν βάση ε, συμβασμού. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα ρόλο κλειδί στην Επιτροπή μας. Βεβαίως ε, θα συζητηθεί κατά κύριο λόγο στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος η έκθεση αυτή, αλλά έχουμε και εμείς ρόλο κλειδί. Γιατί καλό είναι είτε να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία είτε να διακόψουμε νομίζω τις εργασίες μας ε, για να σεβαστούμε και τον κόπο των συναδέλφων. Τώρα, όλα αυτά ξεκίνησαν το 2008 με το πακέτο κλίματος και ενέργειας και πάρα πολύ γρήγορα βεβαίω είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Ε, αποτέλεσμα βεβαίω το οποίο ε, προκάλεσε δισταγμούς σε πολλούς συναδέλφους και πέρασε με μεγάλη ταχύτητα εδώ μέσα στην πρώτη ανάγνωση. Οπότε για το ETS, για το σύστημα εμπορίας, να μην ξανανοίξουμε το πακέτο. Ξέρετε, είχαμε αφήσει εκτός την αεροπορία να προσθέσουμε και την ναυτιλία, αλλά μην ξανανοίξουμε ολόκληρο το πακέτο. Ξέρω πως πολλοί συνάδελφοι ε, ακούνε από τους ε, ψηφοφόρους τους, όλοι βρίσκουν τα benchmarks άδικα, αλλά αφήστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να λειτουργήσει. Επίσης, το 2008 υπήρχε μεγάλη εφορία, είχαμε τις συναυλίες, διασκέψεις, Κοπενχάγη, αλλά ξέρετε τι, που κατέληξαν όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω πως είναι απολύτως απαραίτητο να μην κάθεται στο τραπέζι των παιδιών η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ήταν στην Κοπενχάγη, μιλούσαν οι μεγάλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν με τα παιδιά, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια κλιματική διπλωματία. να μην κοιτάμε από τις κερκίδες, αλλά να διαπραγματευόμαστε και εμείς όταν μιλάμε για μια παγκόσμια κλιματική συμφωνία την οποία χρειαζόμαστε. Γιατί βεβαίω από μόνοι μα δεν θα σώσουμε εμεί τον πλανήτη και αυτό είναι σαφώ. Χρειαζόμαστε τι άλλε μεγάλες χώρες, τι μεγάλες υπήρου. Πρέπει να εξοικονομήσουν και οι άλλοι διοξείδιο του άνθρακα. Είναι σαφές. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Πράγματι, σωστό. Και σωστή η προσέγγιση Τη εισηγήτρια. να έχουμε σαφείς στόχους. Η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνουμε. Να μην παράγεται καν. Και θεωρώ πως ειδικά στον τομέα της κατοικίας μπορούμε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας με την ανακαίνιση των κατοικιών. Αν έχουμε σαφείς κατευθύνσεις για τη διαδρομή αυτή και βεβαίως με το να έχουμε και έναν ορίζοντα προγραμματισμού για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Θεωρώ πως έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό για εξοικονόμηση ε, ε οξυδίου του άνθρακα ε, και πέρα από το ETS και να δημιουργηθούν έτσι πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Για την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα Δεν έχει οριμάσει ακόμα αυτή η τεχνολογία, αλλά δεν πρέπει να την αφήσουμε κατά μέρος. Γιατί έχουμε δύο δυνατότητε. Τρει θα έλεγα μάλλον. Είτε να μην παράγεται διοξείδιο του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω αυτό σημαίνει πως χάλιβα, μετά χημεία, χημική βιομηχανία κτλ. θα φύγουν όλα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω να θέμε αυτό στην Επιτροπή βιομηχανία. Είτε μπορούμε άρα να εκλείουμε στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα ή να ερευνήσουμε τη δέσμευση και αποδίκευση του άνθρακα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, γιατί ξέρετε η αποδοχή είναι, κινείται στο μηδέν για να μιλήσω για τη χώρα μου. Αλλά όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε θα είναι σημαντικά και σημαντικό θα είναι και η επικοινωνία βεβαίω. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μια συζήτηση όπως με τους λαμπτήρες ξέρετε κύριε πρόεδρε άλλοι λένε δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε άλλοι λένε όχι οπότε θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθούμε με την επικοινωνία να εξηγήσουμε γιατί κάνουμε αυτά τα πράγματα. Άρα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα με όλη την νομοθεσία που θα ακολουθήσει από εδώ και μπρος να γίνει μία αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου πολύ σοβαρή και οικονομικού αντικτύπου για οτιδήποτε κάνουμε στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος και αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου για κάθε κράτος μέλος. Τι σημαίνει δηλαδή όταν κάνουμε το α ή το β για όλες τις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν. Αυτό ζητάμε. Ανανεώσιμες πηγές. Ξέρετε, μία μέρα πριν από την καταστροφή στην ε, Ιαπωνία συζητήσαμε με ε, την εισηγήτρια. Εγώ είπα τώρα δεν ε, θα συζητήσουμε την ποινική ενέργεια. Εγώ έχω θέση, είμαι κατά, αλλά θεωρώ πως δεν είναι αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Έχω κάνει και μια πρόταση επίσης για το 2020, αλλά συμφωνούμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια ε, συμβιβαστική γραμμή για τα ποσοστά για το 2030. Ε, για να δώσουμε σε αυτής κατευθύνσεις και στην Κομισιόν για το ποια θα είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθεί και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το δούμε αυτό ουδέτερα από πλευράς τεχνολογίας. Ξέρετε πως η Κίνα εργάζεται με πενταετή σχέδια και εμείς μιλάμε για σχέδια τέσσερα κονταετίας, αλλά τι γίνεται. Μετά από δύο-τρία χρόνια αλλάζει τελείως τεχνολογία. Δεν μπορούμε να πούμε πως θα έχουμε χι αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά από 40 χρόνια. Μπορούμε να θέσουμε ένα πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε και να διατάξουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας. δεν μπορούμε να ορίσουμε ποια τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε καλές επιχειρήσεις, ικανούς μηχανικούς, όπου εάν έχουμε πρακτικούς, λογικούς στόχους θα ε, επιτευχθούν αυτοί. Οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία που θα πρέπει να υιοθετηθεί. Οπότε, συνοψίζοντας, η άποψή μου είναι πως πρέπει όλοι να δεχτούμε να περάσει μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση από το Κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε βεβαίω και μηνύματα που να στείλουμε. Δεν πρέπει να ξανανοίξει το ETS. Και είδατε τι είχε γίνει το 2008. Σαφείς στόχου για ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Είναι σημαντικό και σαφείς στόχοι επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές. Και στο μέλλον, σας παρακαλώ, όχι μόνο οικονομικές και οικολογικές μελέτες αντικτύπου, αλλά και μελέτες του κοινωνικού αντικτύπου. Και όπως σας είπα, ουδέτερη ως προς την τεχνολογία. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πληρέστατη η δουλειά που έκανε και στρατηγική σημασία. Δεν ξέρω τελικά όμως αν θα βρούμε μια καλή λύση μέσα σε μια εβδομάδα. Έχουμε κάνει την πρώτη με τους Κιώδης και έχουμε προγραμματίσει και μια ε, σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, την ενεργειακή απόδοση δεν πρέπει να την εξετάζουμε μόνο σε ένα ε, εργαλείο καταπολέμησης ε, κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο πρόθεσης της ε, ανταγωνιστικότητας. Αυτό φάνηκε και στην ανακοίνωση των δύο επιτρόπων, Hidegord και Ettinger, Επίσης, Πρέπει να το συνδέσουμε αυτό το θέμα με την περιφερειακή πολιτική, με τα διαρθρωτικά ταμεία, με την κοινή γεωργική πολιτική επίσης. Η Ένωση Γεωργών στην Σουηδία ε, υποσχέθηκε μέχρι το 2030 να είναι ουδέτερη ως προς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, δείτε ταυτόχρονα και τις υποσχέσεις ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν τομείς ε, που υπόσχονται να δώσουν τμηματικώς μία λύση για την κοινωνία. Αλλά προφανώς για να δώσουν αυτή τη λύση πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι της λύσης οι ίδιες οι βιομηχανίες. Επίσης θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ των νέων εφευρέσεων, νέων τεχνολογικών ανακαλύψεων και υπέρ της καινοτομίας. Στο δι... Ε, ε, η ΕΠΑ και η Ευρώπη έχουν ένα κοινό πρόγραμμα και μια κοινή ε, εκδήλωση στο Παγκόσμιο Φόρουμ Παραδείγματο χάρη, η εταιρεία μα ε, τι κάνει, ασχολείται με την αιωλική ενέργεια, ε, την ηλιακή ενέργεια. Είναι καταπληκτικά τα αποτελέσματα που έχουν από ε, πλευρά προστασία του περιβάλλοντο, πολέμηση των κλιματικών αλλαγών. αλλά και από τεχνολογικής άποψη. Ισπανία, Ισραήλ και Καλιφόρνια είναι αυτοί που χρησιμοποιούν ήδη αυτή την ε, τεχνολογία. Είναι τεράστιο το δυναμικό. Η Επίτροπος Χέντεγκάρντ ε, ε, έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στο ποσοστό των επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ δηλαδή, 19% η Ευρώπη 28% η Ινδία, πολύ περισσότερο δηλαδή, Νότια Κορέα 35% και 48% για την Κίνα. Οι εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι 1,5% αύξηση, δηλαδή 20,5% συνολικά, άρα το μισό από την Κίνα. Θα πρέπει να δούμε να, ε, δηλαδή πώς συνδυάζουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών με τις προσπάθειες που κάνουμε για την ενεργειακή απόδοση. Ε, και εγώ τους χρειάζεται ευρεία πλειοψηφία. Μάλιστα έχει κέρια σημασία το να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία για να εγκριθεί το κείμενο. Οι στόχοι, καλή και οι στόχοι γιατί έτσι μπορούμε να ε, έχουμε καλύτερε επιδόσει Σε οποιοδήποτε τομέα, εμένα μου αρέσει να έχω στόχου. Όποιο και αν είναι ο τομέα. Ε, και είναι καλή εγχώρη στόχη για την ενεργειακή απόδοση. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες όπως με το πακέτο κατά των κλιματικών αλλαγών. Ήταν τις οι διαπραγματεύσει. αλλά δείτε το δυναμικό που υπάρχει και χρειαζόμαστε ε, στόχου για να δούμε ε, σε τι αποσκοπούμε, τι θα επιτύχουμε ανά χώρα και κυρίως χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς στόχου, διότι για την ενεργειακή απόδοση Ε, θέλουμε αύξηση από το 20% στο 30%. Μόνο αν ασκήσουμε πίεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβουμε νέες προτάσεις που χρειαζόμαστε ούτως ώστε να βαθμίσουμε τα τεχνολογικά πρότυπα, να κάνουμε τις απαιτούμενες ε, επενδύσεις, να ακολουθήσουμε τις κατάλληλες βιομηχανικές πολιτικές. Για το σύστημα εκπομπής ε, ρήπων, το ETS θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, κάποιες βελτιώσεις όντως, αλλά δεν θέλω να ανοίξουμε το κουτί της ε, Πανδώρα σε καμία περίπτωση ε, για το ETS. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να προσθέσουμε πράγματα. Παραδείγματο χάρη, αυτό που κάνουμε τώρα για την ε, αεροπορία, για την ναυτιλία. Από περιβαλλοντική απόψη υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στη Βαλτική θάλασσα, αναβάθμιση των προτύπων των σκαφών που πλέον στην, των πλοίων μάλλον που πλέον στην Βαλτική θάλασσα. Or, fraud. Τώρα στην, ε, για την καταπολέμηση της απάτης. Όταν διαπραγματευτήκαμε το ETS, εγώ είχα υποβάλει σχετικές τροπολογίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως ε, αναθεωρεί, επανέρχεται η Επιτροπή. Μα όλε οι πολιτικέ ομάδε ε, του Κοινοβούλιο είχαν καταθέσει από κοινού την πρόταση στον τελευταίο τριμερή διάλογο ε, και την αποσύραμε όταν ε, διαπραγματευόμασταν με την, το Γάλλο Υπουργό. Θέλουμε μία ρύθμιση όπως αυτή που ισχύει για τα χρηματιστήρια, όχι μόνο. Δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας. Uh, technology τεχνολογική ουδετερότητα. Πολύ σημαντική έννοια επίσης. Τώρα το θέμα των τραπεζών. Αν πρόκειται για αγορά, ε, θα πρέπει να μπορείτε να αποθηκεύετε, να προγραμματίζετε την οικονομία σας. Αυτός είναι ο των επενδύσεων. Οι 10.000 εταιρείε περίπου εμπλέκονται στον τομέα και το κάνουν αυτό. Προγραμματίζουν, υπολογίζουν, παίρνουν τις αποφάσεις τους. Οπότε καλό, καλό είναι, αλλά ε, υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που οφείλουμε να εξετάσουμε περαιτέρω από τη αγοράς. Και πάλι για το ETS, το σύστημα εκπομπή ρήπων, έχουμε δει συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί από τι ΣΥΠΑ δικαιώματα εκπομπή ρήπων για να αποφύγουν κάποιε λειτουργίε τη αγορά. Δηλαδή, αντί να έχουν ανοιχτέ κρατικέ επιδοτήσει για την οικοδόμηση νέων μονάδων ή για να διατηρήσουν παλιέ μονάδε, χορήγησαν ναι, ε, έξτρα δικαιώματα, πρόσθετα δικαιώματα ε, ε, εκπομπής ρήπων. Τρία παραδείγματα μπορώ να κατονομάσω αν θέλετε, όχι τώρα εδώ, μετά κατηδίαν εκτός εθούσης. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μην ανοίξετε το κουτί της Πανδώρας όμως με το ETS γιατί τίποτα δεν πρόκειται να καταφέρουμε και κυρίως όχι μέχρι το 2020. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα ε, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον εισηγητή και του σκιώδεις εισηγητές και σίγουρα θα έχουμε καλέ προτάσει και αρκετά ισχυρή πλειοψηφία στην Ολομέλεια για να αποφύγουμε αυτά που πάθαμε με τα πυρηνικά την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις γιατί ε, κάποια πράγματα δεν έχουν ακουστεί. Όταν μιλάμε για ενεργειακή αποδοτικότητα και έχουμε δεσμευτικούς στόχους και έχουμε μια ημερομηνία αναφοράς, τι έχουμε άρα. Βάζουμε ένα πλαφόν στην οικονομική ανάπτυξη. Μια τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη και ανεξαρτήτως της ενέργειας με την οποία παράγουμε. Έχουμε δηλαδή και τροχοπέδι και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί και να θέλουμε να αναπτυχθούμε με πράσινες μορφές ενέργειας δεν το μπορούμε έτσι. Κάτι άλλο το οποίο ελπίζω να σας προβληματίσει λίγο. Υπάρχουν προγνώσεις ενέργειας από διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται από το 1990 μέχρι το 2030. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο μέχρι το 2030 οπωσδήποτε ο όγκος του διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίω θα πάει από, 40, από 14 ε, σε 40 ε, δισεκατομμύρια τόνους. Ανεξαρτήτως του τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε η Γερμανία θα πάει από το 1 δισεκατομμύριο, θα το μειώσει στα 700 εκατομμύρια τόνους. Κυρίε και κύριοι, είναι ε, ελάχιστο σταγόνα στον ωκεανό σε ο παγκόσμιο πλαίσιο. Σωστό, εντάξει, όσον αφορά και τη μελλοντική τεχνολογία, αλλά πρέπει να δούμε και γιατί μιλάμε εδώ πέρα, το γενικότερο πλαίσιο. Ξέρετε, όταν ε, μιλάμε για το όταν μιλούσαμε στο πρωτόκολλο του Κιώτο για μοίρασμα των βαρών, μιλούσαμε για μοίρασμα των βαρών. Ποια ήταν η μείωση που έγινε. 75% της μείωσης το επομίστηκε η Γερμανία. Και τώρα έχει φτάσει η σειρά των χωρών που είχαν κάποιες παραχωρήσεις. Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη. Εμείς δώσαμε και σκεφτείτε το τι σημαίνει αυτό και για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στο μέλλον. Έχουμε την τρίτη περίοδο εμπορία του συστήματο εμπορία εκπομπών. Είμαστε περήφανοι κτλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τι τιμέ του ρεύματο. 30 με 40% αύξηση στι τιμέ του ρεύματο. Μπορούμε να μιλάμε για διαρροή του άνθρακα κτλ. 30% πάνω. Και τέλο, κάτι άλλο που με ανησυχεί. Τροπολογία κάποιων συναδέλφων για την παράγραφο 2 για να διαγραφεί δηλαδή ότι εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι λόγω των ολοένα αυξανόμενων τιμών ενέργειας φεύγει η βιομηχανία από την Ευρώπη. Δεν θέλουμε καν να το αναγνωρίσουμε. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Σας προσκαλώ να σκεφτείτε τι θα γίνει, να μιλήσετε με ανθρώπους στη Χαλιβουργία, στη βιομηχανία, στη βιομηχανία αλουμινίου φεύγουν οι άνθρωποι, μας εγκαταλείπουν και δεν το συζητάμε καν στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Είναι σκάνδαλο να, να καταθέτουν συνάδελφοι τέτοιες τροπολογίες. Λυπούμε, έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τη μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικές ανησυχίες και κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία ε, κυρίως τώρα που αντιμετωπίζουμε την οικονομική βαθύτατη αυτή κρίση. Η δεσμευτική στόχη για το 2020 είναι ένα σημαντικό εργαλείο και θα μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε ενέργεια μειώνοντας ε, την ε, ενεργειακή μας κατανάλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω Πώς μπορούν οι κυβερνήσεις να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς όρισαν την ενεργειακή απόδοση στο πρωτόκολλο, αλλά ε, ε έχω την εντύπωση ότι ε, δεν μίλωσαν για μείωση της κατανάλωσης, μιλούσαν για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. Είναι ε, δύο πολύ διαφορετικά πράγματα η μείωση κατά 20-25% μέχρι το 2020 είναι ένας μάλλον μη ρεαλιστικός στόχος. Το να επιβάλλουμε ένα τέτοιο στόχο μέσω ε, διοικητικών οδών έχει ως συνέπεια περιορισμούς, επιβολή περιορισμών στην αγορά. Αυτό έχει σημασία αν ε, αυτό που επιδιώκουμε είναι όντω η αύξηση της ενεργειακής ε, απόδοσης και τίποτα παραπάνω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι η μείωση της κατανάλωσης. Θα πρέπει να κάνουμε μετρήσεις κατανάλωσης ανά χώρα ή κατά κεφαλή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πώς η ενεργειακή απόδοση, οι θετικές επιπτώσεις ε, της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης θα μεταφραστούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ενέργεια, ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα οικονομικά αποτελέσματα και με την υποστήριξη της καινοτομίας ε, νομίζω θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε τις εκπομπές, να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να αναβαθμίσουμε ε, την ε, ενεργειακή απόδοση. Συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με το ότι η αύξηση της ε, ενεργειακής απόδοσης ε, κατά 20% θα μας προσέφερε ένα ποσοστό άνω του 20% προς τη μείωση των εκπομπών μπορεί μάλιστα αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση να φτάσουμε και σε μείωση της τάξης του 30% των ε, εκπομπών. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε τον αρισμό της ενεργειακή απόδοση για να είναι ξεκάθαρο για όλους για τι πράγμα μιλάμε. Το ενεργειακό πακέτο και το κλιματικό πακέτο εγκρίθηκε ε, ε, σχεδόν ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη. Ελάχιστε διαστάσεις απόψεων υπήρχαν. Βεβαίω το αναπτυξιακό επίπεδο κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Αυτό νομίζω είναι πρόσκομα σε αυτή την προσπάθεια μείωσης ε, κατά το 20% των εκπομπών στην ε, Πολωνία. Επενδύουμε ε, στην θερμομόνωση των κτηρίων, αποσκοπώντας στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Αν χρησιμοποιήσουμε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ε, τώρα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μείωση του 35%. για τις ε, βιομηχανίες. Τώρα μετεγκαθίστανται ε, εργοστάσια εκτός Ευρώπης και είναι αντίστροφη η τάση. Αν συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τέτοιους περιορισμούς, ενδέχεται να ε, βιώσουμε μια ενεργειακή κρίση στην ε, Ευρώπη. Αυτό μπορεί να συμβεί, είναι... μπορούμε να το φανταστούμε. Κύριος Μιτζάρος, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε από τα λίγα που άκουσα έχω την αίσθηση πως θα είναι αυτή εδώ πέρα η γνωμοδότηση ισορροπημένη. Πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να πω ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες αλλά θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ. Όσον αφορά το πρωτόκολλο του Κιώτο, είχαμε επιτύχει καλά αποτελέσματα στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι εάν παίρνουμε τα πράγματα στα σοβαρά και θέλουμε μέχρι το 2020 να μειώσουμε κατά 20% τις εκπομπές ή και 30%. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και Φαντάζομαι πως μέχρι το 2050 κάποιες χώρες θα έχουν φτάσει αυτό το 90% αλλά αυτό θα είναι επιλεκτικές περιπτώσεις όσον αφορά την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη ε, θα είναι πολύ αβέβαια τα πράγματα δεν θα έχουν επιτύχει το 20% μέχρι το 2020 οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε σε 90 χρόνια ε, μία αύξηση δύο βαθμών. Οπότε θέλω, εντάξει είμαι φυλακτικός, μάλλον θα προτιμούσα να πω ρεαλιστής, ε, γιατί η υπόσχεση που έχουμε κάνει είναι μια εκθετική καμπύλη, δηλαδή στην αρχή πάει εύκολα, αλλά είναι πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα στην αρχή, αλλά μετά γίνεται πάρα πολύ επίπονο αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Όσον αφορά τώρα ενεργητικά και παθητικά μέσα, πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία στον τομέα αυτών, στους στόχους, ενεργητικά μέσα. Τι εννοούμε. Σημαίνει καλύτερο ενεργειακό μείγμα και στη βιομηχανική παραγωγή, να βρούμε νέους δρόμους. Αλλά μετά τη Φουκουσίμα βεβαίως έχουμε μια επανεκτίμηση της ε, πυρηνικής ενέργειας. Θεωρώ όμως αδύνατον να επιτύχουμε τις υποσχέσεις <laughs> μας α, χωρίς ε, πυρηνική ενέργεια. Δεν ε, γίνεται. Πρέπει να συνεννοηθούμε και να ενισχύσουμε την πυρηνική ε, ασφάλεια. Όσον αφορά δε την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως είπαν και οι συναδελφοί, δεν είναι ε, μόνο αυτό το θέμα, να εξοικονομήσουμε ενέργεια, αλλά να δούμε τι γίνεται και στον τομέα της οικοδομής που είναι γύρω στο 40% των εκπομπών και εδώ πέρα αναφέρομαι στα παθητικά σπίτια και πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ ανανεώσιμων πηγών και των οικονομικών μέσων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. Γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υποστορίζουμε τα παθητικά αυτά σπίτια. Ειδικά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτά θεωρώ πως πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παραμένω πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε ε, ολοένα και σαφέστερους στόχους και ολοένα και πιο φιλόδοξους κυρίως ε, στόχους ε, για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020 είναι κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα υλοποιήσουμε. Το στόχο του 17%. Αλλά μπορούμε όμως να ξεπεράσουμε και αυτόν τον στόχο. Υπάρχουν σοβαρές μελέτες, έρευνες που μας λένε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει 30% την μείωση των εκπομπών στο στόχο 2020 για να αναζωογονήσει την οικονομία της. Αυτό σημαίνει τι σημαίνει ότι κατά την επόμενη δεκαετία θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη, εργασία, απασχόληση, θα αυξηθεί το ΕΠ, οι θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις. Σημαίνει ότι θα δώσουμε μια ένεση οξυγόνου στην οικονομία μας που έχει αποδυναμωθεί από την χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά άμα θέλουμε αποφασιστικά να παλέψουμε για το στόχο του 30% πρέπει να ενταχθεί η κλιματική πολιτική σε συντονισμένες φορολογικές και οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσουμε να στοχεύσουμε τις επενδύσεις στις ε, ε, καθαρές ενέργειες low cost. Εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια και την καλό να προχωρήσει προς την υλοποίηση αυτού του νέου στόχου του 30%. Θεωρώ ότι είναι ουσιαστική αυτή η κατεύθυνση στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις επενδύσεις. Γιατί θεωρώ ότι χωρίς ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θα χάσουμε ενέργεια, ε, χρήματα και ανταγωνιστικότητα Οπότε και θα ενθαρρύνουμε μάλλον τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προς την ε, ε, να μετατοπιστούν. Εγώ θεωρώ ότι η Green Economy μετά τη Φουκουσίμα αποτελεί το μέλλον της οικονομίας μας και όχι μόνο γιατί χρειάζεται καθαρή ενέργεια και σίγουρη ενέργεια αλλά επίσης γιατί είναι απαραίτητο αν θέλουμε να εγγυθούμε αηφόρο ανάπτυξη, κυρίως εργασία και απασχόληση. Εγώ πιστεύω ότι μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα και σε αυτήν την κρίση, την οικονομική κρίση, Μόνο ο εγωισμός ορισμένων εθνικών κυβερνήσεων μπορεί να υποτιμήσει αυτές τις θεωρήσεις. Πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει με αίσθηση ευθύνης και κουράγιο αυτόν τον φιλόδοξο αλλά απαραίτητο στόχο. Ευχαριστώ. Ζαντού. Κύριο Ζαντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να εκφραστώ ως ε, σκιώδη εισηγητής. Εγώ ευχαριστώ την Τζορτάνα για τη δουλειά της ε, και για οι προπτικές ε, συζήτησεις που έχουμε είναι πολύ ενθαρρυντικές. Εμείς έχουμε τουλάχιστον τρεις στόχους γύρω από τους οποίους πρέπει να εργαστούμε. Πρώτον, ο στόχος της μείωσης των αερίων, των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πιστεύω ότι θα βρούμε έναν συμβιβασμό γύρω από αυτό. Δεν είναι απλό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Έτσι όπως ε, σήμερα εκφράζεται στην έκθεση η αναφορά στην roadmap του 2050 δεν είναι ακριβής. Αυτό το οποίο λέει ο δικός χάρτης 2050 δεν είναι 20% για να μειώσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα, μειώνοντας και την αναλογία αίτιο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο λέει η roadmap είναι ότι με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχουμε έναν δρόμο. Δεν είναι αναγκαστικά ο καλύτερος, αλλά τουλάχιστον έχουμε έναν αποτελεσματικό δρόμο για να μειώσουμε κατά 25% την οικιακή κατανάλωση και τις οικιακές εκπομπές και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τη συζήτηση. Μετά υπόθηκε από άλλους συναδέλφους ότι συζητήθηκε εξάλλου στην Επίτροπή μας ότι ένας δεσμευτικός στόχος είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και εκπλήσωμαι να ακούω ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι λένε ότι το να εργαστούμε ε, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή για τις οικοδομές ε, είναι κάτι που θα χτυπήσει την ανάπτυξη και την, απασχόληση. Πώς μπορούμε να φανταστούμε σε αυτήν την Επιτροπή να ακούμε ότι το να σταματήσουμε τη σπατάλη είναι κάτι αντιοικονομικό. Και δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε διότι όταν τελικά εμείς παλεύουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας παλεύουμε για την οικονομία, για την πρόοδο, παλεύουμε για την, ε, ε, για, για την ευημερία των πολιτών μας οι οποίοι γονατίζουν από το βάρος ε, των τιμολογίων της ενέργειας. και μπορούμε να ενισχύσουμε τους στόχους μας για την ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να φτιάξουμε ένα πακέτο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και που είναι και ο πρώτος στόχος της όλης συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τελευταίο σημείο. Πιστεύω ότι κυρίως μετά την Φουκουσίμα η συνένεση ή η έλλειψη συνένεσης που έχουμε για την low carbon energy πρέπει να ξαναβγεί στη φόρα. Αυτή η αντίληψη η οποία λέει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνδυασμένες με την πυρηνική ενέργεια και την low carbon energy όλα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο τραπέζι και να τα συζητήσουμε για την για την εξοικονόμηση ενέργειας έλεγε ότι το κείμενο ήταν αρκετά απεσιόδοξο, το συζητήσαμε με την εισηγήτρια ότι το ETS οδήγησε σε μετατοπίσεις επιχειρήσεων. Δεν έχουμε όμως στοιχεία γι' αυτό. Εμείς αυτήν την Επιτροπή καταφέραμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση εξειδικευμένοι και εις βάθος για το ποιοι είναι οι τομείς που ενδυνάμει κινδυνεύουν από την πολιτική για τον, ε, ε, για τον άνθρακα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικά μέσα έχουμε πολύ λιγότερους τομείς από αυτούς που αναφερόμαστε συνήθως ας εργαστούμε γύρω από αυτούς τους τομείς και να μην ξεχνάμε όλους τους τομείς που βγαίνουν κερδισμένοι από αυτή την πρόκληση. Ε, έχουμε πολλούς περισσότερους τομείς ε, στον τομέα και στον τομέα της ε, χωροταξίας που μπορούν να ενισχυθούν και εμείς σταματήσαμε να λέμε ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών πλήττει την οικονομία. Εμείς απασχολούμεθα με εκείνους τους τομείς, τους πιο συγκεκριμένους, που πραγματικά μπορεί να έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι ψέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Αμερικάνοι στην Καλιφόρνια, η Κορέα ε, επενδύουν ε, τεράστια ποσά σε αυτού του είδους την ε, ενέργεια. Εγώ πιστεύω ότι αν τα συζητήσουμε όλα αυτά σε βάθος θα πετύχουμε πολλά πράγματα με τη βοήθεια της εισηγήτριάς μας φυσικά. Η κυρία Χέρτζοκ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην αρχή το σκεφτόμουν να μιλήσω να μην μιλήσω διότι συζητούμε τώρα το σχέδιο ε, για την ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί και προσεκτικοί ταυτόχρονα όταν νομοθετούμε. για να γίνεται ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, τέλος πάντων θα περιοριστώ σε κάποια μόνο σχόλια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Ματές, ότι πρέπει να ε, ομονοήσουμε στο μέτρο το δυνατού στο Κοινοβούλιο, αλλιώς δεν έχει νόημα μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ε, και πιστεύω ότι πρέπει να υπερβούμε το 2020. Υπάρχουν τρεις βασικές προκλήσεις. Πρώτον, η τεχνολογική ε, πρόκληση. Κανείς εδώ μέσα νομίζω δεν θα διαφωνήσει ότι εάν επιθυμούμε να ε, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω μετά το 2020, τότε χρειαζόμαστε ε, σχέδιο για τα ορεκτά καύσιμα, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και για το ΙΤΕΡ. Ένα ε, σφαιρικό σχέδιο. Αλλιώ δεν θα έχουμε ε, καμία δυνατότητα να προχωρήσουμε πέρα το 2020. Δεύτερον, το 2007 το πρόγραμμα προέβλεπε 10 δις για μια δεκαετία. Τελικά το Κοινοβούλιο ψήφισε τα τέσσερα δις, αλλά όχι ως προς, τους, ε, ως προς τις δεσμεύσεις, ως προς τις υποχρεώσεις. Και τώρα βλέπουμε ότι το τελικό κόστος θα είναι 80 δις και ε, είμαστε μόνο το, στο 2011 και εμείς τι έχουμε 4 δις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, ε, αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ μεγάλη χρηματική πρόκληση. Πρέπει να δεσμευτούμε από πλευρά ΙΤΕΡ, να έχουμε τη δέσμευση των Υπουργών Οικονομικών. Ναι, μεν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής ποιος, για ποια χώρα συνιστά αυτό το σχέδιο ε, προτεραιότητα. Για κανέναν. Συζητούμε εδώ τις οικονομικές ανάγκες, ε, προσπαθούμε να έχουμε ομοθυμία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, αλλά είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας, γιατί αυτό δεν συνιστά προτεραιότητα για τα Υπουργεία Οικονομικών των Κράτων Μελών εάν θέλει το Κοινοβούλιο να έχει πυγμή και στένος με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, πρέπει να μεριμνήσουμε πρώτα ότι ε, θα είναι διαθέσιμα τα κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. για να σας εξηγήσω γιατί, αν δεν λειτουργήσουμε μακροπόθεσμα, αν δεν κινηθούν αυτοί που έχουν ε, τα κονδύλια, τι θα κάνουν ε, οι υπόλοιποι. και πώς θα αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό που έχουμε για την ενεργειακή απόδοση, για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν δεν γίνει έτσι. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, τη χώρα, θα πρέπει να αξιοποιήσει την ε, ηλιακή ενέργεια. Προ το παρόν ε, δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Ε, ούτε καν ηλιακού συλλέκτε δεν έχουν τα σπίτια στην Αθήνα. Ε, και νομίζω ότι είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που θα έπρεπε να κάνει τέτοια βήματα. Ε, μόνο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Έτσι θα υλοποιήσουμε το στόχο. Αλλιώ τι είναι, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Κάποιοι θα το υλοποιήσουν, κάποιοι όχι. Αλλά υπάρχουν και χώρε που δεν έχουν τα πετούμενα οικονομικά μέσα για να συνεχίσουν και άρα θα καθυστερήσουν την Ευρώπη. Συγγνώμη, αλλά στην Επιτροπή μα νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια πλειοψηφία ούτω ώστε να κάνουμε κάτι πέρα από το 2020. Δεν μπορείτε να αφήνετε τι χώρε πίσω. Όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε και να υπερβούμε του στόχου του 2020. Ποια είναι τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα. Έχουμε τον προπολογισμό τη Ένωση, τον προπολογισμό των κρατών μελών, το ETS, το σύστημα ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Ε, πολύ ωραία. Αν θέλετε να το τροποποιήσουμε, νομίζω ότι ε, θα έχουμε ελάχιστα αποτελέσματα. Η συγχρηματοδότηση τώρα, πώ χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τη Ένωση, τα εθνικά κονδύλια, αλλά και οι εταιρικέ σχέσει σε δημόσιο ιδιωτικού τομέα και τα project bonds, τα ομόλογα έργων, πώ θα χρησιμοποιηθούν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Προπολογισμών δεν προετοιμάζει έκθεση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή Βιομηχανία να εκδώσει μια ισχυρή έκθεση πρωτοβουλία. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Ε, κατόπιν, έχουμε πάρα πολλέ τροπολογίε. Αν προτίθεστε να προετοιμάσετε προφορικέ ε, τροπολογίε, νομίζω ότι θα ε, συμβάλλατε στο να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Εγώ μία μόνο υπέβαλα, διότι ε, ω προ την πρόκληση για την εφαρμογή, την τρίτη πρόκληση δηλαδή, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα δεν έχουμε λεφτά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, κάνουν κάποιε κινήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ξέρουμε ότι έχουμε 23 εκατομμύρια ΜΜΕ ε, στην Ένωση. Οπότε ε, το 99% δεν θα κάνει τίποτα. Τι θα κάνει το υπόλοιπο 1% των εταιρείων. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομικά μέσα, πρόκειται για αξιοποίηση τοπικού δυναμικού, των δεξιοτήτων, αλλά αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Από τους ε, ηλεκτρολόγους μέχρι τους μηχανικούς. Ε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται σοβαρή οικονομική προσπάθεια και ε, χρειάζεται δέσμευση από πλευρά των εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό χαίρομαι που ο εισηγητής προτίθεται να υιοθετήσει τη σχετική τροπολογία που κατέθεσα. Σας ευχαριστούμε κυρία Χέρζο. Εφτά συναδέλφους έχουμε ακόμα. Θα ήθελα να κλείσει εδώ πέρα ο κατάλογος των ομιλητών συμφωνείτε, ωραία. Και δεύτερον, να σας παρακαλέσω, και μέχρι τώρα άφησα τον καθένα να μιλήσει όσο θέλει, αλλά πρέπει λίγο να επικεντρωθούμε. Δεν λέω δύο λεπτά, αλλά όχι πολύ παραπάνω. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο, παρότι δεν συμφωνώ με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Σύμφωνο απολύτως με αυτό που είπαν πολλοί συνάδελφοι, ότι δηλαδή ε, το έγγραφο αυτό, η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να ταχθεί υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, παραδείγματος χάρη. Συμφωνώ με ε, ε, ο κύριο Ματίας, εγώ είμαι κατά της πυρηνικής ενέργειας, αλλά πιστεύω ότι αυτό το θέμα έχει καταλάβει τεράστια θέση στις ε, τελευταίες συζητήσεις και δεν νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο προς μια καλύτερη απόφαση. Υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, αλλά δεν πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δραστηριότητες για να λύσουμε αυτό το θέμα. Πάντοτε ε, υπάρχουν σοβαρές ε, ε, ανησυχίες όταν τροποποιείται πολύ το περιβάλλον ή όταν έχουμε μια σοβαρή τεχνολογική ανακάλυψη και αυτό σημαδεύει αν θέλετε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε που σχετίζονται με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών σε αντιδιαστόλη με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε συμφωνήσει ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάφορα, διάφορες εκθέσεις όπου ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είναι, είναι εικονική αυτή η αντίφαση. Δηλαδή χρειάζεται προσαρμογή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα όμως το χρειαζόμαστε όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας για να φτάσουμε στο επίπεδο της Κίνας, της Νοτιού Κορέας και άλλων χωρών που επενδύουν πάρα πολλά κονδύλια για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και Εμεί, ε, και πρέπει να προχωρούμε με αυτοπεποίθηση και πεπισμένοι ότι έχουμε δίκιο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ε, και ε, απορώ που υπάρχει αντίσταση ακόμη στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους δεσμευτικούς ε, ε περιβαλλοντικούς στόχους. Μα υπάρχει νομίζω πολιτική ομοθυμία σχετικά με το ότι αν χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο την ενέργεια που ήδη διαθέτουμε θα διευκολύνουμε και την παραγωγή και την κατανομή των ενεργειακών μας πόρων. Είναι ξεκάθαρο ότι για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας ε, θα πρέπει ε, ευθύς αμέσω να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα μας είπατε ότι ε, θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, τεχνικό τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση των τεχνικών στόχων για την ε, μείωση των εκπομπών. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ε, κοιτάξτε, τα κτίρια τα έχουμε καλύψει ήδη τη, για τις ε, οροφές των κτιρίων, εν πάση περιπτώσει, καλύπτουμε εδώ τις μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά επιμέρους στοιχεία μέσα στην έκθεση, πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα για να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δεσμευτικούς στόχους, ε, γιατί χωρίς τους δεσμευτικούς στόχους δεν πρόκειται να σημειώσουμε καμία πρόοδο. Επίσης, θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με πολλά άλλα που είπε ο Ματίας Γκρότε, αλλά ε, συνοψίζοντα θα έλεγα ότι χρειάζονται επενδύσεις. Ε, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα διανομής. Ε, καταλαβαίνετε ότι η ενέργεια από τον τόπο παραγωγής μέχρι τους καταναλωτές ε, σημειώνει πολύ μεγάλες απώλειες. Επίσης πρέπει να επενδύσουμε στα ευφυή δίκτυα τα smart grids και να αποφύγουμε κάθε τρόπο ε, απώλειας ε, των ενεργειακών μας πόρων ε, στον δρόμο από την παραγωγή προς την κατανάλωση. Και ξαναλέω ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις για την πυρηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται εδώ να φαίνεται τέτοια διάσταση απόψεων στη συγκεκριμένη έκθεση πρωτοβουλίας. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο. Και να προσθέσω μόνο το εξής. Πρέπει να συμφιλιώσουμε την κλιματική δράση με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά απαιτεί πιο περίπλοκες λύσεις από ένα στόχο μόνο διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στόχο διοξιδίου του άνθρακα, 20% για το 2020 Έχουμε και οριζόντιες συμφωνίες, π.χ. για την αεροπορία. Άτα την άποψή μου, το να αλλάξουμε τον στόχο σε πιο φιλόδοξο πρέπει να συνδεθεί με μια αποτελεσματική λύση για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών εκείνων που φεύγουν. Για το λόγο αυτό το να έχουμε μια ολιστική οριζόντια λύση θα αυξήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Και αυτό βεβαίως ε, θα βοηθήσει σε μια διεθνή συμφωνία πλαίσιο για το 2010 το τελευταίο. Το τελικό σενάριο διεθνούς συμφωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πλέγμα που θα συνδυάζει τους συνολικούς στόχους αναχώρα με οριζόντιους στόχους όπως έχουμε για την αεροπορία και για τα δάση που επίσης μπορεί να θεωρηθεί οριζόντια συμφωνία. Υπάρχουν ε, επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ε, πώς να συνδυάσουμε αυτές τις προσεγγίσεις. Και τα έχω δει εγώ αυτά για μια παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαρίστως να τα στείλω στους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τη δουλειά που έχω κάνει. Επίσης χαίρομαι γιατί η Κομισιόν στην αρχή ήταν επιφυλακτική και τώρα ε, αγκαλιάζει τη λύση αυτή και ελπίζω να αποτελέσει μέρος της λύσης για να συμφιλειωθεί, να συμβιβαστεί ε, η κλιματική δράση με την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συζητήσω με δύο συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα με την κυρία Χέρτσογκ. Um, Έχετε δίκιο κυρία Χέρτσοκ, πως χρειάζεται να υπάρχει η ευρωπαϊκή ηγεσία. Δεν είναι καλό κάποιοι να φεύγουν πίσω, να προχωράνε και άλλοι να μένουν πίσω στο σταθμό όταν φεύγει το τρένο. Αλλά δεν θα το έλεγα το ερώτημα όπως εσείς. Δηλαδή να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτούς που έχουν μείνει πίσω για να βελτιωθούν. Το πρώτο ερώτημα που θέτω είναι γιατί τα χρήματα της συνοχής δεν χρησιμοποιούνται συστηματικότερα για να προωθεί ενεργειακή αποτελεσματικότητα στο, στα κτίρια που είναι κάτι σχετικά φτηνό. Και στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, που είναι επιτυχή σε αυτό το τομέα, καταρχήν υπήρξε ένα επιχειρηματικό μοντέλο Πρώτα απ' όλα υπήρχε η πολιτική βούληση και μετά δημιουργήθηκε επιχειρηματικό μοντέλο. Οπότε ναι, στη συνοχή, στην αναγκαιότητα να πάμε όλοι μαζί προς τα μπρος, αλλά θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητες προσπάθειες να απαιτηθούν. Δεν μπορεί να ζητάμε συνεχώς νέα λεφτά. Και δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Πίπερ που ε, είπε με αφορά το ζήτημα. Χαίρομαι που επιτέλους ε, ακούγεται και από αυτή την πλευρά το ότι σας αφορά το ζήτημα γιατί αυτό ήταν αγαπητή διατύπωση των πράσινων φονταμεταλιστών μου. Και πρώτον γκρίνια σε υψηλό επίπεδο και δεύτερον μία σπρώμαυρη εικόνα της ε, πραγματικότητας και μια που μιλάμε για τον κύριο Πίπερ, ο κύριος Πίπερ παριστάνει σαν να έπρεπε η Γερμανία λόγω υψηλού ενεργειακού κόστος να γίνει μια ε, βιομηχανική έρημος. 75% του βάρους της μείωσης το φέρει η Γερμανία και δώσαμε. Δηλαδή τι είναι λιγότερο ανταγωνιστική η Γερμανία ή μήπως συμβαίνει το αντίστροφο και έγιναν από τις πιο ανταγωνιστικές χώρες. Εγώ θυμάμαι ήδη πως το BTE είχε υποβάλει μια μελέτη το 2007 που έλεγε πως ε, η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας συνδέεται και συμβιβάζεται με την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε ψηλές τιμές ρεύματος, αλλά αυτό οφείλεται σε ψηλά τέλη διέλευσης. και μην ξεχνάτε πως παίρνουν περισσότερα χρήματα από τις εταιρείες αυτές γιατί δεν υπάρχουν διοικητικές ρυθμίσεις για την τιμή του ρεύματο για τη βιομηχανία αλλά δεν είναι πως ε, η Γαλλία που έχει χαμηλότερες τιμές ρεύματο είναι ισχυρότερη ε, από πλευράς βιομηχανίας έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα της ενέργειας σε σχέση με τη Γαλλία Α, δηλαδή, αν το βλέπαμε μόνο έτσι άσπρο-μαύρο, θα πήγαινε στην Ουκρανία η βιομηχανία που είναι πολύ φτηνή ενέργεια. Ε, δεν είναι έτσι. Όμως, θα ήθελα λοιπόν να βλέπουμε τις πραγματικότητες που μας διδάσκουν πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ φιλόδοξης οικολογικής ε, κατεύθυνσης και καινοτόμων πολιτικής και ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα χωρίς αυτού τους φιλόδοξους ε, καινοτόμου στόχου δεν θα υπάρχει. Ευχαριστώ. Χάση. Thank you very much. Ε. Ευχαριστώ. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, είμαστε στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου το βασικό μας θέμα, δηλαδή τους κλιματικούς στόχους. Ε, έγκριτες επιστημονικές μελέτες ε, καταδεικνύουν ε, πως σε ένα παγκόσμιο θέμα, σύστημα καταμερισμού βάρους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να καταφέρει κάτι περισσότερο από το 30% μέχρι το 2020. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δηλαδή άλλε χώρες στον κόσμο έχουν ε, πολύ καλή επιχειρηματολογία. Δηλαδή ε, ισχυρίζονται ότι αν η Ευρώπη περιορίζεται στο 30% ή και λιγότερο, ή ακόμη και αν είναι πιο φιλόδοξο στόχο, 35-40% παρόλα αυτά δεν ε, αντιστοιχεί στο μερίδιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ούτως ή άλλως ακούγονται τέτοιες φωνές και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα, ε, σε σχέση με το 25% είπε ο συνάδελφος ο Γιάννης Ζαντό, πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τελευταίο δικό χάρτη αναφέρει ότι για να φτάσουμε το 18% το 2005 χρειάζεται να φτάσουμε το 30% εγχωρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ε, τονίσω αυτή την παρατήρηση, διότι αυτό το 25% από πλευράς ε, ε, καλής σχέσης κόστους-οφέλους μπορεί να ε, σημαίνει ότι θα ε, μεταθέτουμε στη συνέχεια τη μείωση των εκπομπών. Δηλαδή, σε εγχώριο επίπεδο σημαίνει ότι αυτή τη δεκαετία ε, θα προχωρήσουμε με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις επόμενες δεκαετίες. Άρα ε, ε, μεταθέτουμε τους στόχους μας ε, στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει μπορούσαμε να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους σε σχέση με αυτό που μας λέει η Επιτροπή το 25% μέχρι το 2020 σε σχέση με την εγχώρια μείωση Πολλές πολιτικές ομάδες ε, ε, τόνισαν πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και θα συμφωνήσω πλήρως με αυτή την άποψη. Σκεφτείτε ποιος είναι ο βέλτιστος ε, δυνατός τρόπος για να ασκήσουμε πίεση για πιο φιλόδοξη πολιτική για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέσα από αυτή την έκθεση σε Ακόμη και η Επιτροπή μιλώντας για αυτή τη βελτίωση του 20% μέχρι το 2020 αναφέρει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί το σωστό δρόμο για να υλοποιήσει το στόχο. Ε, όμως λέει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μείωση του 25% σε εγχώριο επίπεδο δεν είναι κάτι καινούριο, είναι business as usual. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι για να καταφέρουμε το μείον 25% μέχρι το 2020 με εγχώρια μέσα. Τώρα, για να πετύχουμε το 25% της αύξησης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέχρι το 2020, τι σημαίνει ότι θα επιτύχουμε μέχρι το 2020 με χώρια μέσα το 5% της μείωσης. Αν το Κοινοβούλιο θέσει λιγότερο φιλόδοξο στόχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μείον 25% με εγχώρια μέσα μέχρι το 2020, αν πει κάτι λιγότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το στόχο, ε, τότε αυτό δεν συνάδει με τον ε, γενικότερο στόχο μας. Ε, δηλαδή να έχουμε δεσμευτικούς στόχους για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ευχαριστούμε η συνάδελφος Τικάου τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εισηγήσή της. Σχετικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, πολλοί συνάδελφοι είπαν ήδη ότι θα πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια μέσα από πολιτικές αποτελεσματικής ενεργειακής αποτελεσματικότητας στον τομέα των μεταφορών και των κτηρίων. Το μελλοντικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο και εν ώψη της επεξεργασίας του θα πρέπει να διαθέσουμε μεγαλύτερα κονδύλια για την θερμική μόνωση των κτηρίων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών το δυστύχημα της Φουκουσίμα και η συζήτηση για τη χρήση των, της πυρηνικής ενέργειας. Πολύ ωραία. Η επίπτωση ποια είναι ότι στο μέλλον η πυρηνική ενέργεια θα στοιχίζει ακριβότερα από ό,τι σήμερα. Οι χώρες που στο μέλλον ε, που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια στο μέλλον θα πρέπει να δούνε το ενεργειακό τους κοκτέιλ, το ενεργειακό τους μίξ και θα πρέπει να δώσουν περισσότερο χώρο στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι κατεπήγον τα κράτη-μέλη να επανεπεξεργαστούν τα εθνικά τους σχέδια ενεργειακής αποτελεσματικότητας για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μέλλον να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Πυρίλο, ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να... Να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Πρατικό και τους μαθητές από την Καλαβρία. Ο Ματίας είπε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μας ακούνε ακόμη και αν βρίσκονται στη νότια άκρη της Ευρώπης, στην προκειμένη περίπτωση στη νότια Ιταλία. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Ματίας βέβαια είπε πολύ σωστά ότι η καλύτερη οικονομία είναι η ενέργεια, η ενέργεια που δεν καταναλώνουμε. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την ενέργεια στον κόσμο. Και σήμερα το πρωί ακούσαμε νέα όχι και πολύ ευχάριστα από το εργοστάσιο της Φουκουσίμα και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Υπόθηκε από πολλούς προλαλήσαντες συναδέλφους ότι πρέπει να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία διότι θα πρέπει να αποφύγουμε και το επαναλαμβάνω αυτό το οποίο συνέβη στην Ολομέλεια. Δηλαδή ότι ένα κοινοβούλιο δεν καταφέρνει να δώσει ένα μήνυμα για το τι σκέφτεται γύρω από τα πυρηνικά. Εγώ διάβασα αυτό που παρουσίασε η συνάδελφος η συγγήτρια. Πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Φύγονται ένα σωρό σημεία τα οποία φυσικά εγώ δεν θα επαναλάβω αλλά είναι πολύ σημαντικά. Βέβαια θα κάνω και καμιά τροπολογία που πιστεύω ότι μπορεί να βελτιώσει το κείμενο. Μόνο ένα πράγμα θέλω να αναφέρω. Όταν ζητάμε από την Κομισιόν να δώσει προτεραιότητα στις κλιματικές αλλαγές, στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η έρευνα είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Η καινοτομία και η έρευνα δεν περσεύουν ποτέ σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος μιλάει τελευταίος αναγκαστικά επαναλαμβάνει πολλά πράγματα διότι όλοι οι προηγούμενοι κάτι είπαν αλλά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα για το 2030 και το 2050. Εγώ ο ίδιος ήμουνα εισηγητής για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Και επειδή μιλάμε για μεταφορές, εγώ θυμάμαι ότι εκείνο το, το, το μέτρο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση Ήδη λοιπόν ε, με εκείνη την ευκαιρία διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές θέσεις διαφορετικές μεταξύ τους τις οποίες θα πρέπει να ενώσουμε και να καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο συσπηρωτικό για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος και την εξοικονόμηση ενέργειας διότι και τελειώνω αυτή η Επιτροπή ασχολείται κυρίως με βιομηχανία, έρευνα και ενέργεια. Ο κύριος Βέμπερ. Ναι, για να προσεγγίσουμε τον στόχο του 30% εξοικονόμησης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει να δραστηριοποιήσουμε τουλάχιστον τρεις μηχανισμούς που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Φυσικά, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αυτό σημαίνει τεράστιες επενδύσεις και πρέπει, καλά κάνει η Χέρτζοκ που επιμένει σε αυτή τη διάσταση του προβλήματος ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φυσικά και φυσικά μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα σε αυτόν τον τομέα αλλά αν εμείς θέτουμε αυτόν τον στόχο του 30% το 2020 θα πρέπει να προσφύγουμε στην προμήθεια ενέργειας ε, ε, από πυρηνική ε, ενέργεια. Ξέρουμε ότι έχει πολλά από αυτή η ενέργεια, αλλά δεν έχουμε τίποτα καλύτερο και στο βαθμό που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τις ορυκτές και πυρηνικές πηγές ενέργειας, ο αγώνας κατά της θέρμανση, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η εξοικονόμηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος μας υποχρεώνουν να προσφεύγουμε σε αυτού του είδους την παραγωγή ενέργεια διότι ήδη υπάρχουν οι εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται πάνω σε σεισμικά ε, ρήγματα στη Γαλλία για παράδειγμα και που ελέγχονται από το δημόσιο το να βγούμε από την πυρηνική ενέργεια και συμφωνούν και οι πράσινοι. Μια γενιά μας χρειάζονται, 25 με 30 χρόνια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτή την πηγή ενέργειας όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά με απόλυτη ασφάλεια. Και σήμερα σε αυτόν τον τομέα η δημόσια διαχείριση είναι ουσιαστική. Πρέπει να αποφύγουμε ε, να ξεζουμίξουμε τα πυρηνικά εργοστάσια αναζητώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος από αυτά. Χρειάζεται ένας διεθνής έλεγχος, χρειάζεται καταρχήν ευρωπαϊκός έλεγχος, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να ελέγχουν τακτικά αυτές τις εγκαταστάσεις και να υπάρχουν μέσα ε, και στα πλαίσια του παγκόσμιου της οργάνωσης ατομικής ενέργειας να μπορεί να ελέγχει αυτές, αυτές τις εγκαταστάσεις ο συνάδελφος Ράνστορφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Το 87 ε, ο Κέννιντ Αμερικανός ιστορικός ε, εξέδωσε το βιβλίο «Άνοδος ε, και πτώση των μεγάλων αυτοκρατοριών». Είχε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Ε, γιατί ξέρετε η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων ε, πότε συμβαίνει όταν αυτές οι δυνάμεις έχουν υπέρμετρες φιλοδοξίες σε σχέση με τις ικανότητές τους. Και εδώ μιλώ για τις οικονομικές ε, δυνατότητες μιας δύναμης. Αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει σε παρακμή πολλών δυνάμεων, προσπάθησαν να ελέγξουν αλότρια εδάφη, είχαν ε, γενικότερα υπέρμετρε φιλοδοξίες. Πρέπει να αποφύγουμε εμείς αυτό το κίνδυνο. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τις ε, δυνατότητες που έχουμε. Κύριε Μπιουτικόφερ, ε, ισχυριστήκατε ότι η γερμανική οικονομία είναι εύρωστη και έχει καλές επιδόσεις. Έχω μια διαφορετική εντύπωση. Ο κύριος Σρέντερ επέτρεψε 20.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα για, το, για όσους εργάζονται στη βιομηχανία των τεχνολογιών πληροφορικής, κυρίως τον εργάζονται για τη γερμανική αγορά. Από αυτά τα 20.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μόνο τα 1.500 ε, ζητήθηκαν και τελικά υλοποιήθηκε το σχέδιο μόνο για 200 αυτοκίνητα. Ε, οφείλεται αυτό στην κακή φήμη της ε, Γερμανίας, ε, κυρίως στις νέες γενιές, γιατί σε αυτό το τομέα των νέων τεχνολογιών έχει την φήμη σας χώρας η Γερμανία. Ευχαριστώ η κυρία Χέρτσογκ ξανά το λόγο για να επανέλθει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε γιατί με κατονόμασε ο κύριος Μπιουτικόφερ και θα ήθελα να αντιδράσω αν και μάλλον θα βρεθώ στις ουγγρικές εφημερίδες αύριο, θα με λένε προδότη, θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί έχω μια εφταετή ιστορία εδώ μέσα. Εγώ δεν θεωρώ πως είναι κανένας φιλανθρωπικός οργανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε πως στείνονται στην ουρά για φιλανθρωπία τα νέα Το αποδεικνύει αυτό η επταετής πορεία μου, αλλά εξακολουθεί να ισχύει πως εάν θέμε να πάμε πέρα από το 20% δεν επαρκεί να το κάνουν κάποια κράτη-μέλη και 20 να μείνουν πίσω. Γι' αυτό τα νέα κράτη-μέλη δεν ζητάνε φιλανθ... που δεν ζητάνε φιλανθρωπία δεν μπορούν να προσυπογράψουν τους δεσμευτικούς στόχους. Και αν μιλάμε για δεσμευτικούς στόχους πρέπει να αντιμετωπίσετε το ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν τους πόρους να τα επιτύχουν αυτά. Γι' αυτό είμαι κατά του να διασφαλίσουμε με την νομοθεσία αυτή μονοπωλιακά δικαιώματα για τις βιομηχανίες που είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί έχουμε εκλεγεί εδώ πέρα για να εκπροσωπούμε τους λαούς και όχι για τις επιχειρήσεις κάποιων ε, επιχειρήσεων που εντάξει μπορεί να είναι αλλά εγώ δεν έχω εκλεγεί για να δώσω μέσω της νομοθεσίας μονοπωλιακά δικαιώματα σε κανέναν και ήθελα να αντιδράσω γιατί ήταν πολύ προσωπική η αναφορά σας σε εμένα. Αν θυμάστε, εγώ να ζήτησα δραχμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι σε ανταγωνιστική βάση, πείτε μου. Δεν δε, θα ήθελα να, να ξεκινήσω. Τώρα εντάξει θέλει να επανέλθει ο κ. Μπουτικόφερ. Ε, σύντομα όμως. Μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πίπερ που λέει δηλαδή ότι η πολιτική μας οδηγεί στο να μειωθεί πάρα πολύ αν δεν ερημωθεί τελείως η, δική, βιομηχανία στη Γερμανία εσείς μας παρουσιάζετε πως η δική μας η πολιτική είναι λόμπι της γερμανικής βιομηχανίας. Ε, κάπου αυτά τα δύο μεταξύ τους δεν κολλάνε. Ο πρόεδρος. Καλό είναι κάποια στιγμή να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα γιατί και ο κύριος Πίπερ να σας υπενθύμησε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση και νομίζω να πω και κάτι ως πρόεδρος, κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Είναι μια καλή ευκαιρία η έκθεση αυτή να δούμε κάτι το οποίο βέβαια θα είναι δύσκολο, να δούμε τις διαφορετικές πολιτικές θέσεις και να μπορέσουμε να βρούμε μια ησυχία στη συζήτηση γιατί όλοι αυτοί οι στόχοι πιο ψηλά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο μακριά με, ναι, με ανησυχούν και εμένα γιατί έχω την εντύπωση πως ε, δεν, θα επιτύχουμε τίποτα ή ότι βάζουμε πολύ δύσκολους στόχους ή έχουν συνέπειες που δεν τους έχουμε σκεφτεί. Και βιαζόμαστε πάρα πολύ γρήγορα καμιά φορά και θα πρέπει ίσως να τα σκεφτούμε. Και μία δεύτερη φορά αυτά τα πράγματα. Πριν από πολλά χρόνια είχαμε δει το ζήτημα του unbundling της αποδέσμευση σε ένα άλλο θέμα και δεν ε, είδαμε βεβαίως ε, το ζήτημα των μελετών επιπτώσεων. Γιατί αν εμβάθυνε κανείς θα έβλεπε πω δεν είχαμε μπει πάρα πολλές λεπτομέρειε. Οπότε για το θέμα των επιπτώσεων του αντικτύπου, τα έχουμε εξετάσει, το έχουμε δει, ποιε επιπτώσεις έχουν οι αποφάσεις μας. Για κάθε ζήτημα, για κάθε ζήτημα θα έπρεπε νομίζω να γίνει μια συζήτηση έτσι πιο πολύ όσον αφορά τις αρχές αυτών των ε, ζητημάτων που δεν έχει γίνει. Τουλάχιστον για νομοθετικές αποφάσεις όταν λαμβάνουμε να γίνει μια φορά μια ήσυχη συζήτηση και να αξιολογήσουμε να αξιολογήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις εάν έχει γίνει σωστά ή όχι και να γίνουν και πιο εύκολες οι αποφάσεις. Και με συγχωρείτε δηλαδή γιατί Ξέρετε πως ε, δεν μπορώ να μιλήσω πλέον γιατί είμαι πρόεδρος και, και είναι και κουραστικό. Και ο, και ο συνάδελφος που ζήτησε λόγο έχει, έχει τουλάχιστον και αυτός δικαίωμα να μιλήσει. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Λάντσορφ, αν θέλετε. Äh, ε, δεν είναι ευγενικό, θέλω και εγώ να ασκήσω όμως κάποια κριτική σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Έτιγκερ. Τι ήρθε εδώ πέρα χτες ο κύριος Έτιγκερ και ήταν απογοητευτικός. Μόνο λόγια. Δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμος στην Ευρώπη. The roadmap που ανέφερε για τον οδικό χάρτη για το 2020 δεν υπάρχει λέξη για τον άνθρακα. Πώς είναι δυνατόν να, ε, να μην ε, αναφέρεται πλέον στην ενέργεια. Και τώρα οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ε, έρχονται εδώ πέρα και, λέει πώς θα πρέ... και λένε πως και λενε πως θα πρεπει να επαναπεξεργαστούμε τον οδικό χάρτη του 2020 για να μην υπάρχει κανένας ρόλος της πυρηνικής ενέργειας. Απίστευτα πράγματα zu bedauern, dass äh, der alte Kommissar, der ο προηγούμενος επίτροπος, ο κύριος ε, Πίμπαλξ, ε, κακώς εγκατέλειψε αυτή τη θέση. Ήταν πολύ καλύτερος από τον τωρινό επίτροπο, ο πρόεδρος. Ε, το καθένας μπορεί να κάνει τις αξιολογήσεις του, είναι δικαίωμά του, αλλά καλό είναι να γίνει ε, ξέρετε, στην ε, κατάλληλη συζήτηση, γιατί οπωσδήποτε στον ε, οδικό χάρτη θα πρέπει να συζητήσουμε διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια. Και μην ανησυχείτε. Και στη Γερμανία τώρα μιλάνε για ενισχυμένο ρόλο του άνθρακα. Δίας, πρόεδρος μεγάλου γερμανικού κόμματος, ζήτησε νέα εργοστάσια με άνθρακα για να Ε, προχωρήσουμε προς τα μπρος. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως πρέπει να, να τελειώσουμε. Κύριε Λάγκεν, κύριε Λάγκεν ε, επειδή δεν έχετε μιλήσει. Ναι, κοιτάξτε, μόνο για χάρη της αλήθειας. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ, τον οποίο και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, τι ε, έκανε. Τα δύο μοναδικά πυρηνικά εργοστάσια στη χώρα του στην Ιγναλίνα έκλεισαν. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο είναι στην ε, ημερήσια διάταξη και ας ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Γκότε. Και μετά πρέπει να ακούσουμε και την εισηγήτρια και πάμε και παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτη πολύ χρήσιμη έκθεση και πολύ ενδιαφέρουσα ζωηρή συζήτηση γίνεται. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία ζητήματα. Κυρίω ε, πρώτον, σχετικά με τα συμπεράσματα που έχουμε στο σχέδιο έκθεση. Τα καλωσορίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Διότι θεωρούμε ότι είναι χρήσιμε αυτέ οι συστάσει και ότι είναι παρεμφερή σε σχέση με συμπεράσματα και θέματα πολιτική ε, που εξέθεσε και στον οδικό τη χάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, πόσο σημαντικό είναι το στρατηγικό τεχνολογικό σχέδιο, η αξιοποίηση των τεχνολογιών με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Έχουν αυτά ιδιαίτερη βαρύτητα και για την εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων, αλλά και για την ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα ε, στη... και το... για την πρόθεση του μέλλοντο τη ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία για να υπάρξουν δηλαδή νέε αναπτυξιακέ δυνατότητε στον τομέα αυτό. Δεύτερον, η σημασία των επενδύσεων. Και αυτό το τονίζουμε στο δικό χάρτη και αναφέρονται τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα στα συμπεράσματα, μα βεβαίω έχουν ιδιαίτερη σημασία για να τονωθούν οι επενδύσει και να γίνονται σε τεχνολογίε με χαμηλή ε, ε, ε εκπομπή ε, άνθρακα και για να έχουμε ε, μειωμένες ε, εισαγωγές στην Ευρώπη. Συζητώντας τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπολογίσουμε διότι παραδείγματος χάρη διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υψηλό δυναμικό για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στα νέα κράτη-μέλη και για την ερώτηση που μου θέσατε για την κατάσταση στα κράτη-μέλη θα σας απαντούσα ότι εξετάζω συγκεκριμένα τα εθνικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ποιε επενδύσει πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο για να εκπληρώσουμε ολοκληρωθούν οι διάφοροι στόχοι. Τρίτον, σχετικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ρίξατε ιδιαίτερο βάρο στου σχετικού στόχου και είπατε ότι ο δικό χάρτη δεν συνάδει με μακροπρόθεσμου στόχου. Κοιτάξτε. Ε, αυτό με φέρνει στη δεύτερη παρατήρησή μου. Δηλαδή έγιναν διάφοροι πενιγμοί κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, σχετικά με το, το δρόμο, τον, τον προσφορότερο δρόμο πλευρά κόστου κόστου-οφέλου. Δύο πράγματα θα σα πω από αυτού. Πρώτον, αληθεύει ότι όταν ε, συνέταξε τον οδικό τη χάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η μείωση του 25% θα υλοποιηθεί ακολουθώντα αυτό το δρόμο τη ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ε, και γι' αυτό μιλήσαμε για μείωση εγχώρια 20% μέχρι το 2020, δηλαδή το πακέτο όπως ισχύει τώρα ε, και ο δρόμος αυτός ε, σαφέστατα κοστίζει περισσότερο σε σχέση με τη μείωση του 25% ή του 40% σε εγχώριο επίπεδο. Στόχους που θέτουμε δηλαδή μέσα στον οδικό μας χάρτη. Το δεύτερο που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ενισχυμένη δράση για την προώθηση της αποτελεσματικότητας θα μας οδηγήσει σε μείωση του 25% ή και παραπάνω. Ε, επίσης, ακούσαμε διάφορα σχόλια σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ε, βιομηχανιών ε, που, με μεγάλη χρήση ενέργειας, την καταπολέμηση των καταπολεμικών αλλαγών κτλ. Δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποτιμά την διαρροή ε, του άνθρακα. Ε, το έκανε εξάλλου και όταν κλείθη να κάνει αξιολόγηση αντικτύπου για το ενεργειακό πακέτο και στην ενδιάμεση ανακοίνωση το κάναμε και επίση για στον οδικό χάρτη 2005 εξετάζουμε εκ τη σύνεγγυ στο θέμα τη διαρροή άνθρακα. Οπότε στην Ευρώπη έχουμε αναλάβει τα σχετικά μέτρα για τη διαρροή άνθρακα για, την, ε, για το δωρεάν ε, επιμερισμό παραδείγματο χάρη free allocation και θα λέγαμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα αλλά έχουν μειωθεί οι κίνδυνοι σε σχέση με την αρχική μα αποτίμηση πριν από τρία χρόνια για δύο λόγου αυτό πρώτον Άλλες χώρες ε, ε, αναλαμβάνουν μέτρα. Έχουμε τα μέτρα της Κοπενχάγης. Πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε αυτό και ε, φερειπίν βλέπουμε ότι η Κίνα στο πενταετέ σχέδιο εφαρμόζει τη, τη δέσμευση της Κοπενχάγης. Δεύτερον, οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις που κάναμε πριν από τρία χρόνια. Πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ τα μέτρα γιατί είναι πρόσφορα για να αντιμετωπίσουμε τη διαρροή του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ich Ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά ανησυχώ όταν ακούω για πενταετή και δεκαετή πλάνα αλλά δεν ξέρω αυτό μπορεί να οφείλεται στι προσωπικές μου ευαισθησίες. Ε, η συνάδελφος ε, έχει τον, τον λόγο. Ε, ευχαριστώ. Πρόκειται ε, για μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα ε, ζωηρή. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν. Και εναπόθεσαν στους ώμους της υποφαινομένης και των σκιωδών εισηγητών ένα τεράστιο άχθος. Όλοι Ευχόμαστε να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εγγυηθούμε μια σταθερότητα στόχων. Μέχρι το 2020 ζητήθηκαν επαρκείς περιορισμοί για να μπορέσουμε να είμαστε και ρεαλιστές και να έχουμε και μια ισορροπημένη κατάσταση. Το σύστημα ETS πρέπει να παραμείνει όπως έχει, διότι πρέπει να αρχίσει να, να ροντάρει μετά μας είπαμε ότι θα ήταν καλό να συζητήσουμε το όραμά μας για το μετά το 2020. Ο συνάδελφος Ροκ μίλησε για το 2030. Μίλησαμε για την τεχνολογική πρόοδο και λέμε ότι με τα διάφορα μέτρα πρέπει να ενθαρρύνουμε την, στην εξέβρεση νέων τεχνολογιών. Αυτό το οποίο με ενοχλεί κατά τη συζήτηση είναι αυτό το οποίο βγαίνει και ξαναβγαίνει συνέχεια σε γερμανικό επίπεδο. Εύχομαι να έρθουν γρήγορα οι εκλογές στη Γερμανία. Διότι πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε πώς ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενσωματωθεί στις προσπάθειές μας και μετά να προτείνουμε τα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, κάνει, να πράξει ακόμη πολλά πράγματα. Και περιμένουμε εκεί όπου υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας να ε, γίνει και η προσπάθεια. Για τον συνάδελφο Πίπερ και το πρωτόκολλο του Τόκιο, μα όλες οι χώρες ξεπέρασαν τους στόχους του Τόκιο και είχαν καλές επιτυχίες εκτός από τη χώρα μου βέβαια, από τη χώρα την οποία κατοικώ, τη Σλοβενία. Σύμφωνο ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις επενδύσεις. και οι τροπολογίες είναι κάπως αδύναμες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Αν υποβάλλετε προτάσεις ε, θα προσπαθήσω να ενισχύσω το κείμενο και με προφορικές τροπολογίες φυσικά. Παράγραφος 29. Εδώ έχουμε τη θέση της Επιτροπής Ήτρε και λέμε τι πρέπει να κάνουμε για να προσεγγίσουμε και να ξεπεράσουμε τους στόχους μας. Αυτό το τμήμα θα πρέπει να το επανεπεξεργαστούμε με τροπολογίες. Πολλές φορές αναφέρθηκε η ιστορία της συνένεσης. Φυσικά εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε συμπαγείς, να έχουμε τη συνένεση για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να έχουμε, τις, να, έχουμε πλειοψηφία πρώτα στην Επιτροπή μας και μετά στην Ολομέλεια. Πρέπει να βρούμε έναν κοινό δρόμο και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και με και με την εισηγήτρια την κυρία Ετχαούτ για να μπορέσουν αυτές οι δύο εξέσεις να δείχνουν ε, προς μία ενιαία κατεύθυνση. Αν σε επίπεδο περιβάλλοντος και ήτρε καταφέρουμε να βρούμε μία συμφωνία είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μία αξιοπρεπή πλειοψηφία και στην Ολομέλεια η οποία πλειοψηφία θα μας επιτρέψει να έχουμε και μία ενισχυμένη θέση στα θεσμικά μας όργανα. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στα επόμενα. Το πρώτο είναι το υπαριθμόν... Μια στιγμή. Ναι, δημοσιονομικός κανονισμός του προϋπολογισμού. Ο κύριος Οντί είναι ο εισηγητής. Α, όχι, συγγνώμη. Λάθος, λάθος. Κάλβιν, Κάλφιν. Λάθος, λάθος. Κάλφιν και ε, έχει τον λόγο βεβαίως ε, πρώτος. Παρακαλώ λοιπόν. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε ήδη μια φορά το ζήτημα του δημοσιονομικών κανονισμών και το πεδίο ενδιαφέροντος της Επιτροπής μας. Και μιλάμε για τους κανόνες των δαπανών του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού που αφορούν την, ε, τις πολιτικές έρευνας, ε, ανάπτυξης και καινοτομίας και πρέπει να σας πω πως ε, ήταν μακροσκελής η διαδικασία, πολλές φορές ε, πήγαν τα έγγραφα μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και ήρθαν και τώρα το Κοινοβούλιο προετοιμάζεται να ψηφίσει πριν τον Ιούνιο από ό,τι κατάλαβα από την επί της ουσίας, Επιτροπή την Επιτροπή Προπολογισμού και την κυρία Γκρέσλε. Μετά θα έχουμε μια διαδικασία συνδιαλλαγής, ε, αλλά τέλος πάντων τώρα εδώ είμαστε. Το κείμενο το οποίο συζητάμε έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πρώτο κείμενο και την πρώτη επιλογή. Αναφέραμε πολλά ζητήματα που είναι σημαντικά και θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό για να αναφέρουμε τα βασικά ζητήματα. Είχαμε απλοποίηση πρώτα απ' όλα των κανόνων και μιλάμε κυρίως όπως σας είπα για πολιτική έρευνα ανάπτυξης και καινοτομίας. Απλοποίηση είπα να πει πως θέλουμε καλύτερους ορισμούς και σαφέστερους κανόνες στις διάφορες φάσεις ε, εφαρμογή, διαχείριση των κονδυλίων κτλ. Υπήρχε μία ανησυχία που ανέφερε η επιστημονική κοινότητα για την προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα που δύσκολα εφαρμόζεται για τους στόχους της έρευνας και της καινοτομίας και αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε εν μέρη στο κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή, επιτάπητος. Υπήρχε μια ανησυχία για το λεγόμενο ανεκτό κίνδυνο επέλευσης φάλματος και το πώς πρέπει να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο σφάλματος ε, στα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε. Ξέρετε πως το ελεγκτικό συνέδριο το κοιτάει, αλλά όταν μιλάμε για έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να είναι σαφές πως εάν θέμε να ελαχιστοποιήσουμε τα σφάλματα, αυτό σημαίνει να μεγιστοποιήσουμε τη γραφειοκρατία και τους ελέγχους τα λοιπά και κινδυνεύουμε μετά να γίνει αυτό το οποίο λέει η επιστημονική κοινότητα, δηλαδή να χάσει το ενδιαφέρον ε, για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του να αποφεύγουμε τους κινδύνους και να έχουμε λεπτομερείς ε, κινδύνους, ε, ελέγχους με συγχωρείτε, και ε, κάποιας περισσότερης ελευθερίας για την επιστημονική κοινότητα για να μην ασχολείται συνεχώς με τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία αλλά να έχουν μια πρόσβαση στα κονδύλια για να επικεντρωθούν στο επιστημονικό τους έργο. Πρέπει να σας πω πως το κείμενο που έχουμε εδώ πέρα Θα πρότεινα εγώ και κάποιες ε, περαιτέρω διευκρινήσεις, να τονίσουμε το ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη, παραδείγματο χάρη, ο κίνδυνος ε, στον τομέα της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής, στην πολιτική συνοχής και στην έρευνα και ανάπτυξη που θα πρέπει να αξιολογηθεί διαφορετικά ο κίνδυνος στον κάθε τομέα. Όσον αφορά την απλοποίηση, Να σας πω πως ε, το θέμα είναι βεβαίως οι διατάξεις και εκεί πέρα μπορεί να υπέλθει μεγάλη ευλοποίηση, οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάπως ικανοποιητική κατάσταση. Υπάρχει άλλη μια ανησυχία επίσης ε, από την ερευνητική κοινότητα και αφορά βεβαίως κανόνες για την προχρηματοδότηση και βεβαίως υπήρχε μια διαδικασία ενδιαφέρουσα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όσον αφορά τώρα τις ίδιε χρηματοδοτήσεις υπάρχει ένα σαφέστερο ορισμός του τι είναι επιχορήγηση και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πηγαίνει σε μια θετική κατεύθυνση. Επίσης υπάρχει ορισμός των τιμών και τιμέ ορισμένε φορές ε, των βραβείων, με τα οποία δίνονται για την ε, κάτι το οποίο είναι θετικό και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τα κοινότερα μέσα για τη χρηματοδότηση και την προώθηση έρευνας και καινοτομίας και όχι τόσο πολύ τα εξαιρετικά όπως τα βραβεία. Επίσης να αναφερθώ σε δύο έγγραφα τα οποία βρίσκω πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η έκθεση που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συνάδελφος μας κυρία Καρβάλιο που ε, ανέφερε κάποιες πολύ σημαντικές συστάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας καθώς και την ε, τελική έκθεση για το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7 που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2010 και που πάλι δίνει κάποιες περιττέρω διευκρινήσεις που είναι σημαντικές. Ανέφερα πως εγώ θα πρότεινα μια καλύτερη και σαφέστερη μεθοδολογία και ορισμό του τι είναι ο ε, κίνδυνος ε, και θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση αναταμείο και κράτος μέλος. Ε, αυτό σκοπεύω να προτείνω, καθώς και το ότι μπορούμε νομίζω να ζητήσουμε από την Κομισιόν, εάν δούνε μεγάλο υψηλό ποσοστό σφάλματος ε, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, να λάβουν κάποια μέτρα περαιτέρω απλοποίησης ε, ή επανασχεδιασμού του προγράμματος ε, και των διαδικασιών. Αυτές είναι οι βασικές τροπολογίες. Συμπερασματικά μπορώ να πω πως το κείμενο αυτό συνεισφέρει θετικά και θα καταστήσει τους κανόνες ε, χρήσης και χρηματοδότησης ε, απλούστερους. Επίσης υπάρχει βεβαίως η εισαγωγή ενός ανεκτού ποσοστού σφάλματος που πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω και να γίνει πιο ευέλικτος και κάποιο περισσότερο έτσι, βάρος και γραφειοκρατία που υπάρχει στην ερευνητική κοινότητα αποφεύγεται σε αυτό το κείμενο και βεβαίως όταν ψηφίζουμε το κείμενο θα δούμε και τα των εφαρμοστικών διατάξεων. Αυτά θα το δει η Κομισιόν. Εμείς πρέπει να δώσουμε ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συνάδελφο Δελφίν ε, για... Το συνάδελφο, συγγνώμη, Κάλφιν ε, για τις... για την έκθεση του, διότι μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε στη νομική βάση των απλουστευτικών μέτρων ε, που θέλουμε και συγχαίρω και την κυρία Καρβάλιο για την έκθεσή της που λύνει τα, εν μέρη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστημονικοί οργανισμοί ε, για, όλα αυτά. Θα δούμε τι, θα δω τι τροπολογίες θα προτείνω. Τώρα, λεπτομέρειες, παράγραφος 17. Η Επιτροπή λέει πως ε, μαζεύει τις, ε, τα χρέη δηλαδή πώς ε, μετά από συζήτηση ζητάει να τις επιστραφούν τα χρήματα η ανάληψη το, του χρέους ε, πρώτα γινόταν αυτόματα Δηλαδή τα χρέη από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο τα, ε, τα, παίρνανε από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόκειται όμως εδώ για χρέη τα οποία πρέπει να καλύπτονται σε μετρητά και σε κατευθείαν συναλλαγή μεταξύ ε, του λογιστή ε, της ε, Κομισιόν ε, και του Οφιλέτη. Η απλούστευση που θέλουμε, πού θα πάει, σε ποιο τμήμα θα πάει για να πετύχουμε την απλούστευση. Θα βρίσκεται στις βασικές εκτελεστικές διατάξεις της κάθε πολιτικής ή θα έχουμε έναν αυτούσιο κανονισμό. Μου λένε κυρίως όχι δεν θα πρέπει να, ε, να, να αγγίξουμε τις, ε, τη, τη βασική πράξη. Το βασικό είναι να δούμε σε ποιο σημείο θα τοποθετήσουμε αυτή την αλλαγή. Το σημαντικό είναι να τα δούμε όλα αυτά μαζί με την κυρία Καρβάλιο. Δεύτερο, Μήπως ήρθε η ώρα να διαρθρώσουμε τον προπολογισμό μας, το άρθρο 40 του δημοσιονομικού κανονισμού, να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε τον προπολογισμό και να έχουμε την τμήματικοποίηση μεταξύ λειτουργίας και επένδυσης. Δηλαδή η Ένωση εδώ και ορισμένα χρόνια αρχίζει να αναρωτιέται για τον ρόλο της στον τομέα των επενδύσεων. Το είδαμε για τα σχέδια Γαλιλαίο και Ήτερ και για την διάρθρωση του προϋπολογισμού ο οποίος τελικά περιγράφει μόνο τα έσοδα και τα έξοδα και δεν είναι πλέον κατάλληλος ο προϋπολογισμός για τη λογιστική καταγραφή των επενδύσεων σε ε, μεγάλες επενδύσεις που δεν είναι αιτήσιες και πολλές φορές ξεπερνούν και την διάρκεια της μιας δημοσιονομικής προπτικής. Μήπως οι δαπάνες και τα έξοδα θα έπρεπε να ε, κατηγοριοποιούνται μεταξύ λειτουργίας και επένδυσης. Επίσης δεν συζητήσαμε επαρκώς ε, το θέμα με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού στο άρθρο 29. Είναι για το λάθος. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι πολίτες ε, σήμερα θα δεχθούν την ιδέα να έχουμε ένα ανεκτό όριο ε, κινδύνου. Δηλαδή και δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε πάνω σε αυτό το ανεκτό όριο λάθος. Αυτό θα μας, θα, γι' αυτό θα μας κατηγορήσουν μετά. Διότι και το ελεγκτικό συνέδριο έκανε το, τη σύγχυση μεταξύ του ανεκτού ορίου λάθος που είναι μία αρχή ε, της ε, Κομισιόν και την ε, ε, σημαντική αρχή ε, που είναι καθαρά ελεκτικός όρος. Όλα αυτά κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια των αντιευρωπαϊστών και να τα εκμεταλλευτούν. Εγώ είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για, αυτό το, για αυτήν την ιδέα του, του, του λάθους και δεν καταλαβαίνω τώρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ο αριθμός των λαθών ή το ποσό, το μέγεθος του λάθους. Άλλο πράγμα είναι να έχετε 200-300 εκατομμύρια λάθος που μετά το, το, το παίρνει ο τύπος και ε, ε γίνεται πρόβλημα ή έχουμε μετά πολλά λάθη διότι έχουμε πολλούς ε, κανονισμούς ε, πολύπλοκους ε, και ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά, δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο για παράδειγμα για έναν κανονισμό κάνει 180 παληθεύσεις ενώ έχουμε χιλιάδες πληρωμές. Αν ας πούμε ποσοστία τύχης στις 180 ελέγξιμους λογαριασμούς να υπάρχουν λάθη ε, αυτό εννοούμε. Και θα ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κάλβιν. Θα κάνω λίγες παρατηρήσεις και να αφαιρθώ στην τελευταία παρατήρηση του κυρίου Οντί. Θεωρώ την έννοια του ανεκτού κινδύνου επέλευση σφάλματος όχι τόσο απλή. Μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε έτσι παύλο κύκλο. Θυμάμαι πως πέρσι Πέρσι συζητήσαμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και διαπιστώσαμε πως στον τομέα του προγραμματος σε C7 παραδείγματος χάριν είχαμε σοβαρές ε, αποκλίσεις ε, Δηλαδή κάπου το ποσοστό του σφάλματος δεν είναι 2% αλλά φτάνει μέχρι το 5%. Και σε ένα πρέπει να δώσουμε βάση. Πρέπει να προσέξουμε να μην βρεθούμε σε μια κίνηση εκκρεμούς στη φιλοσοφία του προϋπολογισμού. Δηλαδή πρώτα μετά την πτώση της ε, Επιτροπής Σαντέρ είχαμε πολύ μεγάλη αυστηρότητα, τώρα η ποιότητα Οπότε αυτό το οποίο θα πρότεινα για όλους είναι στον κύριο Κάλφιν παραδείγματος χάρη να βρει μηχανισμούς ε, διόρθωσης ε, κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων ακριβώς για να εμποδίσουμε πως ε, η σωστή αυτή πρόθεση ευελιξίας να μην ε, μας κάνει να χάσουμε τον έλεγχο. Ευχαριστώ η κυρία Καρβάλιο. Thank you, Chair. Uh, I would like to... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Our shadow for the... Ευχαριστώ την εισηγητή και τους και τους εισηγητές. Εργάστηκαν πολύ καλά. Στην έκθεση απλούστευσης Υπάρχουν 70 συστάσεις για την απλούστευση του μηχανισμού χρηματοδότησης και των προγραμμάτων χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία. Από τι 70 αυτές συστάσεις, στην ομάδα εργασία εντοπίσαμε Αυτές που μπορούν ε, άμεσα να εφαρμοστούν και κάποιες έχουν εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες άλλες που δεν εφαρμόζονται αλλά δεν χρειάζεται τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και τα έχουμε συμπεριλάβει αυτά στην ενδιάμεση έκθεση του κ. Ντί για το 7ο πρόγραμμα πλαίσια, για την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος και κάποιες ε, που απαιτούν τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Πρέπει να μεριμνήσουμε ότι στην τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού υπάρχουν κάποιες συστάσεις που οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβουμε. Πέντε θα αναλάβω. Μία σημαντική για του ερευνητέ, ε, δηλαδή γενική αποδοχή των ε, λογιστικών πρακτικών για ένα λογικό κόστος, ε, για να χρησιμοποιηθεί ω προ πιστοποίηση, ως μέσο των εθνικών λογαριασμών. Κάτι άλλο χάρση των ε, απαιτήσεων ε, σχετικά με την προχρηματοδότηση. Τρίτον, ε, απλούστευση του μηχανισμού κατά του χρόνου έρευνας, γιατί προς το παρόν ο μηχανισμός αυτός είναι εξαιρετικά περίπλοκος για τους ερευνητές. Τέταρτη σύσταση που ανέφερε και η είναι η χρήση της τιμολόγησης. Πρέπει να διευκρινίσουμε το θέμα κατά την άποψή μου και δεν πρέπει να γενικεύουμε τη χρήση του μηχανισμού των τιμών. Αντίθετα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει η τιμολόγηση, ο προσδιορισμός των τιμών. Τέλος, ε, μείωση της ανάγκης για ελέγχους εξπόστε και αναδρομικών διορθώσεων. Πολύ σημαντικό θέμα για τους ερευνητές μας το ζητούν. Και ε, και συμπεριλαμβάνεται αυτό το στοιχείο, είπαμε, στην ενδιάμεση έκθεση και στις υπόλοιπες συστάσεις. Θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την έκθεση άμεσα με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και με τα χαρές να βοηθήσω τους συναδέλφους, τόσο ώστε οι συστάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στην έκθεση που εκπονούμε για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Κυρία Χέρτσοκ, όχι δεν θέλει πια. Ε, άρα ε, ε, ακούστηκαν όλα σωστά. Οπότε, κύριο ηγητή θέλει πάλι το λόγο. Κύριε Κάλφιν. Α, η Κομισιόν μήπω. Α, δεν είναι κανεί εδώ. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Κάλφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφου που βρήκαν το χρόνο να εξετάσουν ε, το έγγραφο που είναι και δυσανάγνωστο, φίλο να ομολογήσω. Ουσιαστικά συμφωνώ με, τα, με τις βασικές παρατηρήσεις των συναδέλφων. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω τη διατύπωση. Ε, κυρίως αυτό που είπε ο κύριος ε, Οντί για την παράγραφο 117. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε μιλώντας για, ε, για ανεκτό περιθώριο κινδύνου είναι, δεν έχουμε σαφή μεθοδολογία και άρα είναι μια επικίνδυνη στενοπός και πρέπει να προσέξουμε. Ο εισηγητής επιμένει βέβαια να έχουμε το ανοιχτό περιθώριο λάθους, Οπότε αν το έχουμε μέσα στο κείμενο και γι' αυτό έκανα την πρόταση για την ε, παράγραφο 129, χρειαζόμαστε σαφή μεθοδολογία. Πώς θα αποτιμάται αυτός ο κίνδυνος, ποια είναι τα κριτήρια κτλ. κτλ. Διότι Συμφωνώ ότι προ το παρόν δεν υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχει σύγχυση στον τύπο, στο κοινό, ε, σχετικά με το τι εστί ε, ανοιχτό περιθώριο ε, λάθους, ε, ε περιθώριο λάθους. Και αν είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια στο δημοσιονομικό κανονισμό, οπωσδήποτε πρέπει πρωτήτερα να οριστεί επακριβώς. ο κύριος Σιοντή μας μίλησε επίσης για διάκριση ανάμεσα στις επενδύσεις και τη λειτουργία. Δεν ξέρω αν εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε κάτι σχετικό ή όταν θα συζητήσουμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, για τη δομή δηλαδή του προϋπολογισμού. Μαζί με κάποιους συναδέλφους ε, καταθέσαμε και μία τροπολογία βάσει της οποίας θέλουμε ξεχωριστή γραμμή για τα μεγάλα προγράμματα. Είτε πρόκειται για την έρευνα, είτε πρόκειται για άλλους τομείς. Ακριβώς για να μην μπερδευτούμε με τα τρέχοντα προγράμματα της Ένωσης. Αν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε εδώ στο δημοσιονομικό κανονισμό, εντάξει, αλλά πραγματικά είναι θέμα ε, διάρθρωσης δομής του προϋπολογισμού. Ε, that, ε, Mrs. Η κυρία Καρβάλιο τώρα έθεσε διάφορα ζητήματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στα εφαρμοστικά μέτρα, στις εφαρμοστικές διατάξεις ουσιαστικά. Αλλά με τα χαράς αν μπορέσουμε να ενσωματώσουμε κάποια από αυτά τα στοιχεία ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό. Αναμένουμε τις συγκεκριμένες τροπολογίες ε, για τη διατύπωση, αλλά πάντως ε, ακολουθούμε μία και μόνο κατεύθυνση εδώ στην Επιτροπή και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διευκολύνει αυτό το έργο μου. Οπότε τελείωσε εδώ πέρα η συζήτηση αυτή. 3 Μαΐου 12 η ώρα προθεσμία για τροπολογίες. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Περνάμε σημείο 23. Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Ο κύριος Μπιουτικόφερ είναι συγητής. ίδιοι δουλεύουν συνέχεια. Οπότε ο συγητής έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Τα δύο σημαντικότερα θα τα αναφέρω πρώτα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε την εφαρμογή της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 σοβαρά. Γι' αυτό η πρώτη παράγραφος του σχεδίου μου το λέει αυτό με μεγάλη έμφαση χρειάζεται ουσιαστική και συντονισμένη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων για να υλοποιηθούν αυτές οι προτεραιότητες. Η κυρία Χέρτσο που έφυγε είπε θυμίζει πως, ε, μάλλον θα, θα υπενθυμίσω εγώ σήμερα, πως αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να ε, αποδειχθούν τελείως φρούδες εάν δεν τις συνοδεύσουμε με τα απαραίτητα κονδύλια. Και έχουμε άρα ιδιαίτερη ευθύνη και πρέπει να παλέψουμε. Γι' αυτό. Δεύτερον. Και αυτή είναι η παράγραφος παριθμών 6 Πρέπει να δώσουμε βάρος τα διάφορα μεγάλα έργα να μην κολλάνε συνεχώς στον υπολογισμό του σχεδιασμού έρευνας και ανάπτυξης. Είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Έτιγκερ, όπου θετικά κατά την άποψή μου είπε ο κύριος Έτιγκερ πως πράγματι δεν είναι δυνατόν το ίτερ να κολλάει συνεχώς ε, με τις υποχρεώσεις της χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας. Αντιθέτως πρέπει να τα δούμε αυτά ως δύο ξεχωριστά πράγματα ανεξαρτήτως του πόσο ικανοποιημένος είναι κανείς ή δεν είναι από το ίτερ. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μεγάλα έργα και το ίτερ είναι ένα μόνο, το Γαλιλαίο είναι ένα άλλο να υφίστανται συνεχώς αυτή την αυθόρμητη τάση να τρώνε από τις υφιστάμενες πολιτικές μας α, προτεραιότητες. Οπότε θα πρέπει στον προϋπολογισμό να γίνουν τα ανάλογα τρίτη παρατήρηση. Θεωρώ, δεν χρειάζεται πώς να σας το εξηγήσω σε αυτή την επιτροπή, πως ε, οι προϋποθέσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία πρέπει να βελτιωθούν εάν είναι να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Ε, τα έχω πει αυτά. Ε, Ειδικά στη δεύτερη παράγραφο και το τρίτο. το τρίτο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα των προοπτικών των μικρών επιχειρήσεων. Για να τονίσουμε πως το ΣΥΠ στα διάφορα υποπρογράμματα του εξαιρετικά αποτελεσματικό ε, σε δύο πτυχές. Πρώτον γιατί έχει υψηλό ποσοστό κονδυλίων που φτάνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι θετικό κριτήριο και δεύτερον γιατί υπάρχει υψηλή αποτελεσματικότητα στη διοίκηση των κονδυλίων. Άρα προκύπτει για εμένα πως πρέπει να το ενισχύσουμε ανεξαρτήτως ε, του τι θα γίνει με το ερευνητικό πλαίσιο και το πώς λέγεται αυτό. Δεν θα λέγεται πρόγραμμα πλαίσιο 7, αλλά ανεξαρτήτως του ονόματος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις θετικές εμπειρίες με το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να τον ισχύσουμε και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πως υπάρχουν άλλοι σε αυτό το κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας που είπαν πως ε, δεν πρέπει να παίρνουμε τόσο σοβαρά τα προγράμματα αλλά να μπουν όλα σε ένα όνομα. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Τα προγράμματα αυτά τα οποία αποδεικνύονται αποτελεσματικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τα ενισχύσουμε. Η κυρία Χέρτσοκ. Είμαι και με αυτή την ιδιότητα θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικό γιατί παίρνει τόσο πολύ στα σοβαρά τον προϋπολογισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Επιτροπή με πάσα σοβαρότητα διαδραματίζει το ρόλο της στον τομέα αυτό. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλους τους οικονομολόγους για να φτιάχνουν ε, σχέδια για να υλοποιήσουμε εμείς τους στόχους 2020. Ε, ένα γενικό σχόλιο, τρία μάλλον. Γιατί ο προπολογισμό 2012 πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων 2020. Τι θα ξυπνήσουμε το 2020 ξαφνικά και θα πούμε ουτς δεν τα καταφέραμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ε, είναι μια προϊούσα διαδικασία και άρα ο προπολογισμό ε, του 12 πρέπει να ευθυγραμμιστεί με του στόχου του 20. Δεύτερον, ο προπολογισμό 2012, αν θέλετε, είναι μία αίθουσα αναμονής ε, για το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα λόμπι. Ε, οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι μα για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και σίγουρα ο προπολογισμό του 2012 θα πρέπει να ακολουθεί στην ίδια κατεύθυνση. Είναι κέρια σημασία σε αυτό και νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανεί εδώ μέσα, ούτε ο συγητή ούτε οι συγητέ. Ε, λοιπόν, αυτή, αυτός ο προπολογισμό του 12 ε, και να αναφερθώ τώρα εν συντομία στα δύο τελευταία χρόνια του προηγούμενου πλαισίου, γιατί αναλάβαμε πάρα πολλέ δεσμεύσει και τώρα πρέπει να εκταμιευθούν τα χρήματα και πρέπει εμείς να πιέσουμε. Γιατί αλλιώς πλήττεται η αξιοπιστία της Ένωσης αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση και πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Ε, θα συμφωνήσω με σχεδόν όλα τα σημεία που ανέφερε ο εισηγητή. Θέλω όμω να τονίσω ότι υποστηρίζω πλήρω, αμέριστα, ε, το να ζητήσουμε ενεργό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, αυτό είναι ο μονόδρομος για να ακολουθήσουμε το στόχο που αναφέραμε στο προηγούμενο σημείο, δηλαδή να υπάρχει ομοφωνία, ούτω ώστε να μην ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο να είναι ένα βιομηχανικό, επιχειρηματικό και όχι μόνο οικονομικό εξάμεινο. Αυτό πρέπει να, αυτή πρέπει να είναι η μόνιμη ποδόσμα στο μέλλον και ευχαριστώ τον κύριο Πιτικόφερ που ε, συμπερίλαβε αυτό το στοιχείο και πρέπει να ακολουθήσουν οι πληρωμέ, οι εκταμιεύσει, ένα αυτό και δεύτερο με τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα Μιλήσανε για το ίτερ, υπάρχει και το Γαλιλαίο και διάφορα άλλα. Πρέπει να πιέζουμε, δεν πρέπει να ε, εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες. Κάτι άλλο που λέγαμε χτες για την Ένωση της Καινοτομίας. Διευρύναμε το πεδίο της ε, καινοτομίας, πολλαπλασιάσαμε το πεδίο, δηλαδή από την υψηλή τεχνολογία, την αιχμή τη τεχνολογίας, περάσαμε στον τομέα των υπηρεσιών, ε, της κοινωνία των ε, πολιτών, την καινοτομία τη βάλαμε παντού δηλαδή. Όμω, δεν αυξήσαμε τα κονδύλια. Τι σημαίνει αυτό. Τα διαθέσιμα ε, χρήματα για τα τωρινά προγράμματα θα μειωθούν. Άρα θα πρέπει να ε, επιδιώξουμε αύξηση, γιατί αν συνεχίσουμε σε να διευρύνουμε το πεδίο, ε, απαραίτητα αυτόματα θα μειωθούν τα κονδύλια που διαθέτουμε σε κάθε πρόγραμμα. Και ναι. νομίζω ότι... Τι άλλο έχω να προσθέσω. Α, ναι, ήρθε η ώρα να προετοιμάσουμε τα πιλωτικά προγράμματα. Αν ε, προετοιμάσουμε κάποια τέτοια πιλωτικά προγράμματα, θα σημειώσουμε επιτυχία στις προηγούμενες δεσμεύσεις μας, αλλά και στις επόμενες. Θα υποβάλουμε μια τροπολογία, ελπίζω να συμφωνήσουν οι πράσινοι, βάσει της οποίας θα θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ανακαινισμένων ε, ανοιχτών κτηρίων όπου οι πολίτες μπορούν να δουν απτά αποτελέσματα της προσπάθειας που κάνουμε για την αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ελπίζω αυτά, αυτή η οίκη να είναι ε, σκόρπια ανά την Ευρώπη, ούτως ώστε οι επισκέπτες να πηγαίνουν, να αναβοσβήνουν τα φώτα, ε, να δοκιμάζουμε τα έπιπλα των φιών αυτών κτηρίων. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να υπάρξει αφοσίωση και δέσμευση. Χαρητήρια και πάλι στον εισηγήτη. Kollege Saudakas als next. Saudakas. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ε, μιλήσω αγγλικά για να είμαι σύντομο. not so ε, for... Ε, δεν έχουν απομείνει και πολλά να πω, γιατί συμφωνώ πλήρω σχεδόν με όσα είπε η ο εισηγητής ε, και ο κ. Χέρτσοκ γιατί είναι βεβαίως τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευρώπη 2020, αηφόρος ενέργεια, εφαρμογή προγράμματος πλαισίου, Ε, νόμος περί μικρών επιχειρήσεων λοιπά. Αλλά από την άλλη μεριά του μικροφόνου θα ήθελα να πω και εγώ να προσθέσω πως ε, στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης εγώ θα ανέφερα κάποιες λέξεις κλειδιά όπως ε, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, υποδομές στρατηγικού σχεδίου τεχνολογι... ενεργειακής τεχνολογίας. Γιατί, γιατί τον αναφέρουμε αυτές τους τομείς κλειδιά και άλλες λέξεις κλειδιά. Σωστό είναι, αλλά μετά το να παραλείψουμε άλλες ε, είναι ένα αρνητικό μήνυμα. Ότι δηλαδή οι άλλες που έχουμε παραλείψει δεν είναι τόσο σημαντικές. Οπότε θα ήθελα να ξαναμπούν αυτά τα θέματα τα οποία έχουν παραλυφθεί. Δεν ξέρω βεβαίω. Ε, όταν έρθουν τα πραγματικά νούμερα θα μιλήσουμε με πραγματικά νούμερα. Και τέλος για αυτό το περίφημο άρθρο 6 της γνωμοδότησης που πιστεύω θα συζητήσουμε να προσθέσω κι εγώ μια διαφορετική πτυχή ε, ε, γιατί είναι το πώς θα ξοδευτούν αυτά τα πολλά λεφτά. Αλλά βλέπετε, αναφέρουμε το Ίτερ, αναφέρουμε το Γαλιλαίο, αλλά από την άλλη, ήδη εδώ στην Ευρώπη, εδώ και πολλά χρόνια, πολύ καιρό, ξοδεύουμε πολλά λεφτά. will not be Άρα εάν αυτά τα έργα δεν θα είναι επιτυχία, θα χάσουμε τα λεφτά που ξοδεύσαμε. Πρέπει να μας ενδιαφέρει λοιπόν η επιτυχία αυτών των έργων Αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε. Οπότε όταν έρθουν τα πραγματικά νούμερα θα ξέρουμε και τι έχει αλλάξει στη γνωμοδότηση της Κομισιόν σε σχέση με την περσινή θέση και τι θα αλλάξει στη θέση του Συμβουλίου και θα διαμορφώσουμε και εμείς τη δική μας θέση για την ε, πλήρη ε, ευθύνη που έχουμε έναντι αυτών των έργων. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπιουτικόφερ, θέλετε να επανέλθετε. Ε, σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, α, ε, μου είπε η συγγήτρια της ε, κύριας εκθέσεως στην Επιτροπή Προϋπολογισμού πως είναι διατεθειμένη να λάβει υπόψη αυτά τα οποία είπαμε. Βεβαίως, δεύτερον, Ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις ε, των ε, δύο συναδέλφων. Έχετε δίκιο, κυρία Χέρτσογκ. Πρέπει, όπως το κάνατε πέρσι, να προετοιμάσουμε αυτό το PAPP και θα το κάνω αυτό και ελπίζω βεβαίως φέτος να έχουμε ένα πιο σύντομο κατάλογο για να συμφωνήσουμε σε περισσότερα πράγματα. Για αυτό το οποίο λέτε εσείς κύριε Τάκας έχετε δίκιο. Είμαι κάπως πιο επιφυλακτικός γιατί πιστεύω πως δεν είναι δυνατόν το σχέδιο αυτό με τόσο έτσι υποθετικούς στόχους να χρηματοδοτήσουμε κάτι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό γίνεται μόνο εάν υπάρχει κάτι ουσιαστικό στον προϋπολογισμό. και δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την πραγματικότητα και να μην δημιουργούμε ε, φρούδες ελπίδες για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το 2012. Αλλά αλλιώς συμφωνώ, πρέπει να μπουν και άλλες λέξεις κλειδιά. ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 Μαΐου, προθεσμία για τροπολογία. και ερχόμαστε στο σημείο 24 ε, της εβδομάδας, δύο οργανικός διάλογος για τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο Τζάιλς Τσίτσεστερ ε, είναι ο πεσταλμένος μας και τον παρακαλέσαμε να υποβάλει μια έκθεση. Γιατί ξέρετε πως αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρο το Κοινοβούλιο, όχι μόνο για την Επιτροπή μας και χαίρομαι για το ότι ε, ανήκει στην ομάδα αυτή ο Giles και θα ακούσουμε μια ενδιάμεση έκθεση. Έχετε λοιπόν το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μήπω έπρεπε να γίνει και κλεισμένο των θηρών η συνεδρία. Θα προσελκύσω το ενδιαφέρον. Θα θέλω να μάθω τι γίνεται πίσω από τι κλειστέ τι πόρτε. Μπόρεσα να τα καταφέρω να με διορίσει η ομάδα μου εισηγητή για το θέμα. Ε, αυτό το έκανα διότι είναι ε, για διάφορους οργανισμούς αυτό σαφές, ε, σαφώς υπέρ των συμφερόντων της Επιτροπής μας και με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα ούτως ή άλλως, Γιατί, όπως και το ενίσα. Θα ήθελα να σας δώσω το, το ιστορικό υπόβαθρο. Το τελευταίο σημείο δεν είναι πρόεδρε, οπότε θα προσπαθήσω να μακρηγορήσω εξαιρετικά ναι. Αλλά τόσο πάντα με βαρεθείτε, κάντε με ένα νόημα να σταματήσω. Uh, Πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία, το Μάρτιο του 2009, όταν τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν να δρομολογήσουν ένα διαθεσμικό διάλογο για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, με στόχο να αξιολογήσουν την ε, επιστάμενη κατάσταση και να βρουν ένα κοινό παρονόμαστη για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Συστάθηκε η ομάδα εργασίας λοιπόν και τη ανέθεσαν να εξετάσει διάφορα σημεία κλειδιά που πρότειναν ε, τα θεσμικά όργανα που συμμετείχαν ε, στο διάλογο. Μεταξύ άλλων, ο ρόλο των οργανισμών στο γενικότερο θεσμικό ε, περιβάλλον της Ένωσης, ε, η συγκρότηση, η δομή και η λειτουργία των οργανισμών αυτών, η χρηματοδότησή τους, ο δημοσιονομικός έλεγχος και τα θέματα διαχείρισης. Η ομάδα εργασίας τώρα του Κοινοβουλίου ε, αποτελείται από έξι μέλη. Η κυρία Χάουγκ από τους σοσιαλιστές και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών προεδρεύει. Η κυρία Γκρέσλε, επίσης από την Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου Προπολογισμών συμμετέχει από το ΕΛΚ, το ξέρετε αυτό βέβαια. Η κυρία Γένσεν από τους Φιλελευθέρους, εγώ από τους Συντηρητικούς, η κυρία Λάμπερτ από τους Πρασίνους και ο κύριος Σμιτ από ε, το EFD. Παρότι οφείλω να ομολογήσω ότι λάμπει δια της απουσίας του στις συνεδριάσεις το Κοινοβούλιο σε μηνιαία βάση περίπου συνεδριάζουμε, διότι είναι ογκοδέστατο το πακέτο των ε, πληροφοριών ε, που μας έχουν δώσει για το ιστορικό της υπόθεσης από την Γραμμάτια ε, και ο Επίτροπος Σεφκοβίτς από πλευρές Επιτροπής ηγείται της προσπάθειας. Υπάρχει και τεχνική ομάδα βεβαίως προσωπικό που εργάζεται άοκνα για να προετοιμάσει τις συνεδριάσεις. Τέσσερα σημεία μας απασχολούν, κατάσταση, τα κρίσιμα προβλήματα, οι πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και τρόποι εφαρμογής αυτών των λύσεων. Τα δύο τελευταία μου φαίνονται πολύ φιλόδοξα σε σχέση με την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει εξετάζουμε το θέμα. Η ίδρυση των οργανισμών, η έδρα τους, ο ρόλος της χώρας που υποδέχει τον οργανισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο, διορισμός των διευθυντών, κοινή διοικητική υποστήριξη, υλικοτεχνική υποστήριξη. Θα μπω σε κάποιες λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα αλλά ας πω αρχικά ότι συζητούμε αν επιθυμούμε να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση. Γιατί αυξήθηκε ο αριθμό των οργανισμών τα τελευταία χρόνια και όχι, δεν πρόκειται για ad hoc οργανισμούς. Ε, ε, ε, έγιναν προτάσεις από διάφορα κράτη-μέλη εξετάζοντας την κατάσταση από διαφορετικές οπτικές γωνίε, όπως διαπίστωσα, γιατί ασχολήθηκα και με το θέμα ε, καθότι ήμουν εισηγητή για το ΕΝΙΣΑ. Μέχρι πρόσφατα τα κράτη-μέλη με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα διατήρησαν τη διακριτική τους ευχαίρεια για να προσδιορίζουν ε, την έδρα των ε, οργανισμών αυτών. Αυτό άλλαξε βέβαια λόγω του ότι το Κοινοβούλιο είναι πλάκι στις συνολικότερες αποφάσεις ε, κάποιων οικονομικών θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει αυξημένες αρμοδιότητες τώρα στη διαδικασία προσδιορισμού ε, της έδρας των οργανισμών, διότι και όπως πρότεινε εξάλλου εγώ προσωπικά στο Συμβούλιο, με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει σε σχέση με διάφορους οργανισμούς. Αλλάζω συνήθεια καπέλα, ιδιότητες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είμαι και ε, στην ομάδα εργασία, είμαι και εισηγητής για τον ΕΝΙΣΑ. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο ΕΝΙΣΑ προκύπτει ως ε, φοβερό παράδειγμα για ε, ότι δηλαδή ε, έχουν ε, προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα για την έδρα του ΕΝΙΣΑ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λοιπόν, ας αρχίσω με τη συγκρότηση, την ίδρυση των οργανισμών. Ο... Συζητούμε αν πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια ε, για τον προσδιορισμό της έδρας. Προσπαθούμε λοιπόν να θεσπίσουμε ενιαία κριτήρια σε σχέση με τον ε, ε, διορισμό υπηρεσιακού διευθυντή μέχρι ότου να διοριστεί ο κανονικός διευθυντής, ο μόνιμος διευθυντής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να φέρει την ευθύνη μέχρι ότου να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ο οργανισμός και ε, μέχρι να δρομολογηθεί η διαδικασία για το διορισμό του ε, μόνιμου διευθυντή και δεν σας ξαφνιάζει ότι το Συμβούλιο αντιδρά σε αυτή την αρμοδιότητα τη Επιτροπή. Τώρα, ο ρόλο της χώρα που υποδέχεται τον οργανισμό, το θέμα της έδρα. είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα από τα δυσχερέστερα σημεία προ διαπραγμάτευση. Τα κράτη-μέλη μεταξύ του ε, αποφασίζουν πού θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα νέο οργανισμό ε, το το γετούγο, όπως λέμε στα γαλλικά, δηλαδή το παζάρεμα για να το πω κοινά, είναι το βασικό χαρακτηριστικό ε, στις, ε, στο διάλογο για τον προσδιορισμό της έδρας. γίνεται μια μοιρασιά ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ένα κράτος μέλος έχει τρεις οργανισμούς, πολύ γενναιόδωρο, μερίδιο έχει πάρει. Και υποτίθεται ότι υπάρχει ένας διακανονισμός ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και τον οργανισμό σχετικά με τις υποδομές που θα προσφέρει η χώρα υποδοχής. Αυτό σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Προς το παρόν να συζητούμε αν πρέπει να υπάρχει απέτηση καν για κοινά κριτήρια σχετικά με τα, τις παροχές ε, που οφείλει να εξασφαλίσει η χώρα υποδοχής. Ε, και όπως σας είπα γίνεται και κάποια συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία που θα συνυπολογίζονται για να αποφασίσουμε τον τόπο εγκατάστασης του οργανισμού και άλλα συναφή ζητήματα, ε, διότι αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, τους εμπειρογνώμονες ε, να μετικήσουν σε ένα απόμακρο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους ανάγκες που δεν ναι, σχετίζονται μόνο με έναν αξιοπρεπή μισθό. Ε, οι οργανισμοί αυτοί κατόπιν έχουν ε, μια δομή, ένα διοικητικό συμβούλιο και γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, πόσο μεγάλα πρέπει να είναι, πώς πρέπει να επιλέγονται τα μέλη τους, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ως προς τη δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Συζητεί δηλαδή αν πρέπει να έχει δικαίωμα άρνηση κυρίας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μέσα στα Διοικητικά Συμβούλια των ε, Εκτελεστικών Οργανισμών. Συνεχίζεται η συζήτηση διότι ε, κάποιοι από αυτούς τους οργανισμούς έχουν και διοικητικά συμβούλια ε, και τεχνικές ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, που είναι τεράστιες ως προς τον αριθμό ε, των μελών σε σχέση με το συνολικότερο αριθμό το, του προσωπικού δηλαδή των οργανισμών. Το επόμενο σημείο που συζητούμε είναι το θέμα των κοινών κριτηρίων για το διορισμό του διευθυντή του οργανισμού. Ε, είναι ε, ρόλος κλειδί αυτός του διευθυντή ε, του οργανισμού γιατί ο ή διευθυντής είναι το σημείο επαφής ανάμεσα στον οργανισμό και το διοικητικό του συμβούλιο Αφενό και αφετέρου τα κράτη-μέλη και το κοινοβούλιο και συζητείται το θέμα των διαδικασιών επιλογής και διορισμού ε, των διευθύντων. Μέχρι στιγμής υπάρχει τάση να διορίζεται ο διευθυντής και κατόπιν ο ε, διάδοχος, ο υποψήφιος, έρχεται στην αρμόδια επιτροπή για μια ανταλλαγή απόψεων. Εμεί πιέζουμε για να αυξηθεί ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε αν ε, θα τα καταφέρουμε στις διαπραγματεύσεις τελικά. Πάντως, το Συμβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει ότι το Κοινοβούλιο μετά την έναρξη τη θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι ένας μηχανισμός ε, ασφαλείας αν θέλετε. Είμαστε ε, το μόνο αιρετό σώμα στην Ένωση και θα μπορούσαμε να επικουρήσουμε το Συμβούλιο για να αποφευθούν οι δυσκολίες. Uh, Αυτά για το διορισμό των διευθυντών. Ε, τώρα, με σε διάφορες συσκέψεις προσπαθούμε ε, να ε, καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις. Δεν το έχουμε καταφέρει όμως προς το παρόν, ναι, Πρόεδρε. Συνεχίζεται το, συνεχίζονται ο διάλογος και ελπίζουμε ότι το ευθυνόπορο θα καταφέρουμε να βρούμε κάποιες λύσεις και να τις υποβάλουμε Το θέμα ποιο είναι, ακόμη και να καταφέρουμε μελλοντικά να έχουμε ένα κοινό σετ κριτηρίων, έχουμε ήδη 32 οργανισμούς διαφόρων ειδών, οπότε αναδρομικά το να τροποποιήσουμε ε, τον τρόπο λειτουργίας τους ε, συνιστά, πώς να το πω, μεγάλη πρόκληση, μεγάλη δυσκολία ε, ή μπορεί να είναι και αδύνατη αυτή η τροποποίηση. Πιθανώ. Δεν μπορεί να είναι κάτι αδύνατο βέβαια. Πιθανώ, αλλά τέλο πάντων είναι αυτή η κατάσταση, όπως σας την περιέγραψα, ε, δεν ξέρω αν ε, υπάρχουν ερωτήσεις ή αν θέλουν οι γενναίοι συνάδελφοι που έμειναν εδώ μέχρι το τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης να μου θέσουν κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και μπορούσατε ίσως να μας βοηθήσετε στέλνοντας ένα κατάλογο στους συναδέλφους ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, πού βρίσκονται, τι κονδύλια έχουν και πόσο προσωπικό. Δεν είναι αναγκαίο όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ένας τέτοιος κατάλογος θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί υποθέτω πως έτσι εύκολα στείνουμε μια τέτοια υπηρεσία, αλλά μετά σε τι εξελίσσεται κάτι τέτοιο και τι γίνεται με τα λεφτά και αν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά νομίζω είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δημοκρατικός έλεγχος, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι κοστίζουν και αν υπάρχει μόνο αυτός ο δρόμος ή υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Και συμφωνώ βεβαίως με την εκτίμησή σου πως πλέον υπάρχει ένας αυτοματισμός που δεν ε, είναι πάντα υπέρ της ουσίας. Η Ενίσια ήταν ένα παράδειγμα μόνο. Ε, γιατί μόλις ξεκινήσει μια συζήτηση γίνεται πολύ συναισθηματική μετά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που μας ενημέρωσες. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το άκουσα πότε θα έχουμε αποτελέσματα συγκεκριμένα. για να έχουμε κι εμείς κάποιο ρόλο κοινοβούλιο. Αν ε, δεν έχει να πει κάποιο άλλο συνάλφο, κάτι νομίζω μπορεί ο Τζάιλ να απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως ο στόχος είναι να ολοκληρώσουμε το έργο μας μέχρι το τέλος του έτους, του 2011. Και σκοπεύουμε να έχουμε και περαιτέρω συναντήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου και τριμερείς ε, και εσωτερικές για το σκοπό αυτό. Αλλά όπως ξέρετε άλλο η επιθυμία και άλλο η πραγματικότητα. Αλλά η πρόθεση, πάση περιπτώσει, είναι αυτή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κανείς δεν θέλει το λόγο, οπότε μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ και υπενθυμίζω στους εναπομείναντες πως μπορούμε να συναντηθούμε στις 12.30 γιατί θεωρώ σημαντικό να έχουμε ένα σωστό αποχαιρετισμό του επικεφαλής της γραμματείας γιατί ήταν μια ξαφνική απόφαση και εγώ θεωρώ σωστό να ήταν κάποιοι συνάδελφοι εδώ ελπίζω να μην φύγετε όλοι και δεν ξέρω ίσως και κάποιοι από αυτούς που έφυγαν να ξανάρθουν σας ευχαριστώ πολύ Giles θέσετε κάτι άλλο παρακαλώ ναι η εκδήλωση θα γίνει εδώ, έξω. Α, ωραία, ευχαριστώ.